εργασία ε, στο πρόγραμμα του τρίου αυτού και εύχομαι κάθε επιτυχία στην Πολωνική Προεδρία που ακολουθεί. Ευχαριστώ κύριε Γκέρι. Ολοκληρώθηκε τη συζήτηση και περνούμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης. Πρόκειται για την έκθεση του συναδέλφου Ντέσσα, κοινή γεωργική πολιτική με χρονικό ορίστο το 2020, αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή του φυσικού πόρου και το έδαφο, έγγραφο Α7-0202 κάθετο 2011. Και παρακαλώ πρώτο τον συνάδελφο και εισηγητή κύριο Ντέσ να λάβει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Πριν από 50 χρόνια, το 1961, ξεκίνησα την κατάρτισή μου ως γεωργό. Έκτοτε η κοινή γεωργική πολιτική είναι πάντα στο πλευρό μου, με συνοδεύει. Αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας ενοποίησης Ευρωπαϊκής Ένωσης με πολύ σημαντικές δαπάνες και καθήκον. Καθήκον πρώτιστο ήταν η εξασφάλιση επιστηστικής αυτονομίας για την ευρωπαϊκή κοινότητα. Λίγο αργότερα προέκυψαν πλεονάσματα τροφίμων στην Ευρώπη με μια κατάσταση που επαναλαμβανόταν διαρκώς και νέες μεταρρυθμίσεις δηλαδή να την αντιμετωπίσουμε βρεθήκαμε τώρα στην κατάσταση να συζητούμε τη νέα διαμόρφωση της χειρουργικής πολιτικής από το 2013 και μέχρι το 2020. Ως εισηγητής λοιπόν Χαίρομαι ιδιαίτερως γιατί καταφέραμε οι πολιτικέ ομάδε να καταλήξουμε σε μια συνένεση, σε μια συμβαστική λύση, έστω και αν δεν ελήφθησαν υπόψη όλε οι αποκλίνουσες απόψει, που επέτρεψε την έγκριση σε επίπεδο της Επιτροπής μας τη εκθέσεω. Σαφές μήνυμα δηλαδή προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πω η Γεωργική Επιτροπή είναι ε, έχει σαφή εικόνα για το πώ πρέπει να διαμορφωθεί η κοινή γεωργική πολιτική έω το 2020. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταβάλει προσπάθεια για να πάρει το πράσινο φως και να φέρει και την υπογραφή του Κοινοβουλίου η κοινή πολιτική από το 2013 και μετά, όπως προβλέπουν και οι συνθήκες. Οι συνάδελφοι Μπάλλοντε Κάστρο, σκιώδεις συγητές, συντονιστές, ήταν πάντα πρόθυμοι για συνεργασία. Με στήριξαν με τις προτάσεις τους. Ευχαριστώ ιδιαίτερως τη γραμματεία της Επιτροπής των πολιτικών ομάδων, τους συνεργάτες και τους δικούς μου προσωπικούς συνεργάτες. Τώρα για την έκθεση θα ήθελα να πω ότι η επιστηστική ασφάλεια αποτελεί κύριο στόχο πάντα της κυρίας γεωργικής πολιτικής, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρέπει η, η γεωργία, η κοινή γεωργική πολιτική να είναι βιώσιμη, αεφόρος και ανταγωνιστική. Χρειάζεται λοιπόν παραγωγή υψηλής ποιότητας τροφίμων, και ανάπτυξη αηφόρων μορφών ενέργειας. Οι δύο πυλώνες της ε, ΚΑΠ θα πρέπει να διατηρηθούν και για την προσεχή περίοδο θα πρέπει να εξασφαλιστούν μέσα προστασίας των γεωργών. Στην έκθεση διατυπώνουμε σαφώς το αίτημα και εδώ υποστηρίζουμε τις προτάσεις του Επιτρόπου στην προσεχή περίοδο να διατηρηθούν οι ενισχύσεις της κοινή γεωργικής πολιτικής στα τωρινά επίπεδα. Στις προτάσεις του κυρίου Μπαρόσου, εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω ότι θα πρέπει ο δεύτερος πυλώνας να περικοπεί μαζικά. Πιστεύω ότι όλες οι πολιτικές ομάδες έχουμε αντίθετη γνώμη στην υπόθεση αυτή. Σημαντικό καθήκον επίσης παραμένει η απλούστευση της κοινή πολιτικής. Αποτελεί κεντρικό αίτημα της συμβιβαστικής πρότασης την οποία έχουμε καταλήξει. Ισότιμη κατανομή μεταξύ των κρατών μελών επίσης ζητούμε. Επίσης λέμε ότι θα πρέπει να εξασφαλιστούν ισότιμες συνθήκες πρόσβασης στον ανταγωνισμό. Οι α, τιμές αναφοράς, ιστορικές τιμές αναφοράς ως προς τις ε, ε, επιδοτήσεις με βάση την ε, έκταση ε, θα πρέπει να διατηρηθούν. Η αρχή της επικουρικότητας και η στήριξη από τα κράτη-μέλη του μικρότερου, ε, του μικρότερου ισχύ ε, αγρότη θα πρέπει να διαφυλαχτεί επίσης πρόσθετα συστήματα ενισχύσεων θα πρέπει να μην οδηγήσουν ε, σε ε, απώλεια του στόχου της διαφύλαξης και της περιβαλλοντικής λειτουργίας της γεωργίας αλλά και της στήριξη των κανόνων. Έτσι λοιπόν όπως έλεγα έχουμε μια έκθεση την οποία ελπίζω θα μπορέσουν οι συνάδελφοι στο σύνολό τους να υποστηρίξουν όσο δυνατόν περισσότεροι και που δίνει σαφή μηνύματα και κατευθύνσει για την κοινή γεωργική πολιτική. Η δική μου πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα την υποστηρίξει πάντως με μεγάλη πλειοψηφία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντές, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Επίτροπος κ. Τσόλος. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Σίγητα, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η έκθεση αυτή κατατίθεται σε κρίσιμη χρονική στιγμή όταν δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το μέλημα της προετοιμασία των μεθοδικών προτάσεων που προβλέπεται να υποβληθούν στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο προ εξετάσεις τον Οκτώβριο. Ευχαριστώ τον εισηγητή κύριο Ντές. για το, την εργασία του τους τελευταίους μήνες, αλλά και την Επιτροπή Γεωργικής Πολιτικής για τις συζητήσεις, τον πλούτο των συζητήσεων και τις ιδέες που προσέφερα κατά τη διάρκεια αυτών και που μα βοήθησαν πολύ στη δικασία αυτή προετοιμασία τη μεταρρύθμιση και τη πολιτική. Πολλά στοιχεία τη εκθέσεω συγκλίνουν ε, με το όραμα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το όραμα που θέλησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει προ με την ανακοίνωση για τη μεταρρύθμιση τη κοινωνική γεωργική πολιτική που παρουσιάστηκε στα τέλη του 2010. Ιδιαίτερα δεν αναφέρομαι στο ζήτημα της επιστημιστικής ασφάλειας ως κύριο στόχο τη κοινή γεωργική πολιτική, αλλά και στη σημασία τη διαφύλαξη των δύο πυλώνων τη κοινή γεωργική πολιτική που ανέφερε και ο κύριος Δε. Επίση, την αναγνώριση τη αναγκαιότητας για πιο πράσινη κοινή γεωργική πολιτική και προσανατολισμό προς την ενσωμάτωση και τη ε, χρηστής διαχείρισης των φυσικών πόρων. Επίσης αναφέρομαι σε μια πιο δίκαιη κατανομή των πόρων της κοινωνικής πολιτική μεταξύ των Ευρωπαίων γεωργών. Και αναφέρομαι επίσης στην αναγκαιότητα να υπάρχει ένας, ε, ε, ένας προϋπολογισμός ο οποίος είναι στο επίπεδο που απαιτούν οι συνθήκες και οι ανάγκες. Επίσης, ανώτατα όρια στις άμεσες πληρωμές όπως αναφέρατε εσείς. Εγώ θα ήθελα για το θέμα αυτό να σημειώσω, να υπογραμμίσω τη σημαντική συμβολή αρκετών μεγάλων ε, εκμεταλλεύσεων στην απασχόληση στην Ήπεθρο. Άρα λοιπόν θα ληφθεί αυτό το γεγονός υπόψη ω προς τον προσδιορισμό του ανώτατου επίπεδου ε, στην ενίσχυση, την οικονομική άμεση οικονομική ενίσχυση των ε, γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Ο πρώτος πυλώνας σε συνδυασμό με μια ενισχυμένη πολιτική ανάπτυξη Ήπεθρου αποτελούν σταθμοί στόχους για την αντιμετώπιση και τον, για την ανταπόκριση στις κλιματικές αλλαγές αλλά και την ε, σαφή ε, εξυπηρέτηση των στόχων της στρατηγικής του 2020. Με ικανοποίηση σημειώνω το γεγονός ότι η έκθεση ζητεί πιο στενή διασύνδεση των άμεσων πληρωμών, άμεσων ενισχύσεων και της διαφύλαξης των φυσικών πόρων. Και στόχος δικός μου είναι ε, να παρουσιάσω ένα πλέγμα προτάσεων με στόχο ακριβώς την εξυπηρέτηση των στόχων μας η αποσύνδεση των άμεσων πληρωμών είναι για μένα πολύ σημαντικός ε, στόχος ε, γιατί απεδείχθη η σημασία της. Αλλά όπως λέτε και στην εκθεσή, της, σας συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και σε ορισμένους τομείς για λόγους ε, ε, οικονομικούς, οικολογικούς ή κοινωνικούς τομείς, δηλαδή που είναι πιο αδύναμοι σε αυτά τα τρία πεδία, θα πρέπει να δοθούν ακόμη και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Αυτές θα έχουν σημαντικό ρόλο για τη διαφύλαξη της ζωτικότητας των διαφόρων περιοχών, πρόκληση δηλαδή που ιδιαίτερα, ιδιαίτερη σημασία έχει στις περιοχές που έχουν πληγεί από διάφορα φυσικά, φυσικά προβλήματα και καταστροφές. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στόχο έχει να προσφέρει και ενίσχυση στο συμπληρωματικό εισόδημα οποιοδήποτε χάρη στο δεύτερο πυλώνα ε, εγκαθίσταται και αναπτύσσει δραστηριότητα σε ζώνες με φυσικό μειονέκτημα. Εσείς αναφέρεστε στην ιδέα αυτή με την προσθήκη ενός ε, συμπληρώματος σχετικού στον πρώτο πυλώνα μια συνιστόσα δηλαδή. Και εγώ προτείνω ένα ειδικό καθεστώ για υποστήριξη και ενίσχυση των μικρότερων εκμεταλλεύσεων με να δυνατόν απλοποίηση των διοικητικών ε, και γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων για τις μικρές αυτές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες ταυτόχρονα θα μπορούσαν ε, να ε, στηριχθούν αποφασιστικά στο πλαίσιο και του δεύτερου πυλώνα, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης έτσι ώστε να μπορέσουν να αναλάβουν ένα ρόλο πιο ουσιαστικό και αποφασιστικό και για την υπεθρο αλλά και ως προς την οικονομική του δραστηριότητα για να είναι πιο αποδοτικές αλλά και πιο ανταγωνιστικές ο γεωργός που παραμένει σε δραστηριότητα θα είναι ο μόνος αποδέκτης αυτών των ενισχύσεων και πιστεύω ότι σε αυτό συμφωνούμε και εσείς και εγώ προς τα οράματά μας για την κοινή κυριολογική πολιτική ε, για το μέλλον. Και έτσι πιστεύω θα μπορέσουμε να βρούμε έναν ορισμό εφαρμόσιμο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα λαμβάνει βέβαια υπόψη και σε ορισμενα ορισμένα κράτη-μέλη συνθήκες. Ε, η πρόταση σχετικά με τις συνθήκες αγοράς ε, μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Η ενίσχυση ικανότητα διαχείριση και τη δυνατότητα λήψη αποφάσεων των ε, παραγωγών αλλά και των οργανώσεών του, η διαμόρφωση των τιμών και άλλα μέτρα σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων είναι μέτρα και ιδέε τι οποίε δεσμεύομαι να μελετήσω πολύ προσεκτικά στην ανάλυση των επιπτώσεων, κατόπιν τι οποίε ε, δεσμεύομαι να καταθέσω πολύ συγκεκριμένε προτάσει. Επίση, συμμερίζομαι τι αναλύσει ω προ την ενίσχυση και την ανάπτυξη μέτρων ενίσχυση τη υπαίθρου και την αναγκαιότητα τα μέτρα αυτά να ανταποκρίνονται πιο αποφασιστικά στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, την ανάγκη εξυπηρέτηση βιοπικιλότητα και τη φύλαξη των φυσικών πόρων. Ο μελλοντικό δεύτερο πυλώνα τη κοινωνική πολιτική θα πρέπει να ανταποκρίνεται όχι μόνο σε αυτέ τι ε, προκλήσει, αλλά και σε μια γεωργία τη γνώση που μπορεί να οικοδομήσει το μέλλον τη κατά τρόπο βιώσιμο με ανταγωνιστικότητα και οικολογικά. Σα διαβεβαιώνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σύνολό της, συλλογικό όργανο και ο Πρόεδρο Μπαρόσο υποστηρίζουν το δεύτερο αυτό πυλώνα ω στοιχείο ουσιαστικό και ζωτικό της κοινωνικής πολιτική. Επίση, για του νέου γεωργούς συμφωνώ με τι παρατηρήσει ότι θα πρέπει να προσφέρετε ένα ευρύ φάσμα μέτρων στήριξη που θα ανταποκρίνονται στι ανάγκε του. Και θα ήθελα να επισημάνω και τα μέτρα που θα ενσωματωθούν στον πρώτο πυλώνα τη κοινωνική πολιτική για του νέου γεωργού. Σημειώνω επίση ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μπορούν στο μέλλον να προσδιορίζουν υποπρογράμματα, θεματικά μέτρα δηλαδή, τα οποία θα απευθύνονται προς το νέο ε, γεωργό και θα το καθιστούν προτεραιότητα για το κράτος μέλος. Κατάρτιση, επαγγελματική εξειδίκευση, υπηρεσίες ενημέρωσης, ε, επενδύσεις για τον εξυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση της εκμετάλλευσης. Όπως άλλωστε και εσείς υπενθυμίζετε, στην εκθεσή σας η πολιτική μας απαιτεί και επαρκείς πόρου έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στι προκλήσει του μέλλοντο. Αυτή τη στιγμή είμαστε εν αναμονή τη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το μελλοντικό πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο θα παρουσιαστεί μέχρι το τέλη Ιουνίου, η οποία πρόταση μάλλον, και Βάσει αυτό τη προτάσεις θα προβούμε στην ανάλυση επιπτώσεων και τι προτάσει για τη χρηματοδότηση και τη ζωική πολιτική μέχρι το φθηνό που σα είπα νωρίτερα. Ευχαριστώ πολύ για την έκθεση και είμαι στη για να δώσω απαντήσει στι ερωτήσει ε, εν αναμονή μια πολύ επικοδομητική συζήτηση. Είμαι βέβαιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. Ακολουθούν τώρα οι ομιλητέ από τι συναρμόδιε επιτροπέ. Ο κύριο Αρσένη πρώτα απ' όλα για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, συζητάμε σήμερα για τη νέα ΚΑΠ. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί που κάνουν την κριτική ότι η κοινή μα αγροτική πολιτική έχει οδηγήσει σε περιβαλλοντική υποβάθμιση, αλλά και έχει απειλήσει και απειλεί, κυρίω τα απειλή στο παρελθόν, ε, τι αναπτυσσόμενε χώρε με πολλού τρόπου, ιδίω τη γεωργία του και την ανάπτυξή του έχουν δίκιο όσοι κάνουν αυτή την κριτική. Όμω έχουν άδικο όσοι ζητάνε ότι πρέπει να μειωθούν οι πόροι για την κοινή μα αγροτική πολιτική. Η κοινή μα αγροτική πολιτική δεν είναι μια πολιτική για τη γεωργία μόνο. Είναι μια πολιτική, ε, είναι ένα εργαλείο αναδιανομή πόρων από τι ευρωπαϊκέ πόλει στην ευρωπαϊκή Ήπεθρο. Είναι οι Ευρωπαίοι πολίτε τη ευρωπαϊκή Ήπεθρου που φροντίζουν τα δάση μα, τα ποτάμια μα, τι λίμνε μα, μα δίνουν τροφή ε, καθαρό οξυγόνο ε, και νερό. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα να αλλάξουν τα κοσκήμενα, ναι. Όμως θα πρέπει να, αν είμαστε σοβαροί θα πρέπει να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση για την αγροτική μας πολιτική, για μια κοινή αγροτική πολιτική πιο δίκαιη, πιο αποτελεσματική και πιο βιώσιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Αρσένη για την Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, και Τροφίμων ε, Κάντενμπαχ για ένα λεπτό. με κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες ε, και κύριοι, εάν ρωτήσει κανείς τους Ευρωπαίους τι περιμένουν από την ευρωπαϊκή πολιτική, έχουμε την ποιότητα ζωής και όριο όπως η υγεία και το περιβάλλον και αυτά σχετίζονται με τη γεωργική πολιτική η οποία θα πρέπει να έρθει στο ύψος αυτών των προσδοκιών των Ευρωπαίων. Και θεωρώ πως η συνεισφορά της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος ε, και ε, Τροφίμων θεωρώ πως είναι ακριβώς να δώσουμε αυτό το οποίο θέλουν οι Ευρωπαίοι. Υγιή τρόφιμα τα οποία παράγονται με βιοπικιλότητα και από πλευράς βιολογικής και από πλευράς μεθόδων παραγωγής. Θα πρέπει να διατηρηθεί ο ζωτικός χώρος και να φροντίσουμε βεβαίως την φύση, ο ζωτικός χώρος επίσης την Ήπεθρο να αναπτυχθεί και να μην ε, καταλήξει να είναι η φτωχή περιοχή της Ευρώπης. Θα πρέπει να έχουμε μια πολιτική γεωργίας που θα φροντίζει όλες τις περιφέρειες. Χρειαζόμαστε γι' αυτό λεφτά, χρειαζόμαστε τα λεφτά σωστά και με δίκαιη κατανομή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο συνάδελφος από την επόμενη επιτροπή δυστυχώς ε, δεν έχει έρθει. Έχει έρθει ο κύριος Σικέρης και από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη. Ε, να πάρα το λόγο. Ε, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, σημαντικό είναι για εμάς η γεωργία σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον να είναι ίσχυρη. Χρειαζόμαστε μια νέα γεωργική πολιτική με ανταγωνιστικότητα στις διεθνείς ε, αγορές και θα πρέπει να έχουν και ένα εισόδημα. Η γεωργή, η ποιότητα των προϊόντων θα πρέπει να διασφαλιστεί, η ανάπτυξη της και βεβαίως το περιβάλλον. Όλα αυτά πρέπει να αποτελέσουν μέλημά μας και βεβαίως θα είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχουν διαφανή κριτήρια για την στήριξη των γεωργών. Και βεβαίως θα πρέπει να δούμε και τους ε, ιστορικούς ε, εταίρους μας ε, στην Ήπεθρο να στηρίξουμε τις οικογενειακές γεωργικές επιχειρήσεις και σβήνει το μικρόφωνο του κυρίου Σικέρσκη περνάμε στους ομιλητές εξ των ομάδων πρώτα απ' όλα Νταντέν για δύο λεπτά Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι Επιτρέψτε μου καταρχάς να χαιρετήσω την ε, δουλειά του συναδέλφου και εισηγητή Άλμπερτες των εισηγητών, των ε, συντονιστών και σκιωδών εισηγητών για ένα έργο, για ένα αποτέλεσμα πολύ ισορροπημένο και πολύ σημαντικό που θα ψηφίσουμε αύριο. Έξι μήνε περίπου μετά του προσανατολισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ΚΑΠ μετά το 2013 με την έκρηξη του κ. Λάινεν, η, Επιτροπή Γεωργία αποφάσισε να στηριχθεί στο έργο αυτό. Με τι ε, συστάσει τη ΔΕΕ στι 18 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπη έπραξε το ίδιο. Και έτσι η, Ευρωπα... Επιτροπή Γεωργία ομόφωνα σχεδόν εγκρίνει την έκθεσή τη και επικυρώνει την μεταστροφή που ζητούμε για την κοινή γεωργική πολιτική και τα επόμενα χρόνια. Δεν παράγουν ένα απλό εμπόρευμα οι γεωργοί μας, δεν είναι απλώς προϊόν δηλαδή εμπορεύσιμο αυτό που παράγει ο γεωργός. Παράγει τροφή, τρόφιμα για τα 500 εκατομμύρια των συμπολιτών μας. Ταυτόχρονα με τη δουλειά του όμως συμβάλλει και στην ε, ε, σύντηση ολόκληρου του κόσμου. Πρόκειται για μια όχι σημειολογική μόνο επιλογή, αλλά φιλοσοφική από πλευράς μας. Η έκθεση του Αλμπερντές προβαίνει σε μια θετική αξιολόγηση της συμβολής γεωργίας και στο περιβάλλον και στην οικολογία και έτσι ζητεί την άρση των πολλές φορές βαριών γραφειοκρατικών συνθήκων που επιβάλλει η ευρωπαϊκή ή η εθνική νομοθεσία πολλές φορές. Και έτσι με μέσα νέα και με σταδιακή εξέλιξη των μέτρων ε, ορίζει την παγκόσμια προσέγγιση και το όραμα της ΚΑΠ αλλά και την εξυπηρέτηση των παγκοσμίων αγκών. Και την ώρα που ξεκινάει το μεγάλο συνέδριο για τη ρύθμιση των πρώτων υλών και δι των γεωργικών υλών στο Παρίσι, η ε, έκθεση αυτή παίρνει μια διαφορετική σημασία και αποδεικνύεται ότι η δική μας δουλειά δεν είναι μεμονωμένη και αποκομμένη από τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά επιτρέπει να δοθούν απαντήσεις παγκόσμιες σε οικουμενικές προκλήσεις όπω την έκθεση Λάιρεν, όπω την έκθεση Γκαρίγκα για τι δημοσιονομικέ προοπτικέ. Αύριο θα έχουμε να συζητήσουμε και τη διατήρηση του γεωργικού προπολογισμού για την περίοδο 2013-2020. Ξέρω ότι έχουμε πολλή δουλειά στην υπόθεση αυτή, αλλά όταν έχουμε να, να λαμβάνουμε επιλογέ, όταν έχουμε να κάνουμε επιλογέ. Ευχαριστώ κύριε Ντόντσε. Είχατε δύο λεπτά μόνο χρόνο. Και ακολουθεί ο κύριο Λουφόλ πάλι για δύο λεπτά. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Πίτροπε. Κύριε Σιγητά. Ο Μισελ Ταντζά εξάντλησε το χρόνο του και έτσι του κλείσε το μικρόφωνο, αλλά ήταν στο σημείο που μας εξηγήσε πόσο σημαντική είναι αυτή η έκθεση για την παγκόσμια ε, οικονομία και είναι όντως πάρα πολύ σημαντική. Η έκθεση αυτή, η δουλειά της Επιτροπής δείχνει και αποδεικνύει ότι χρειάζεται μια κοινή γεωργική πολιτική που θα εξασφαλίσει την ε, επιστημιστική ασφάλεια στην Ευρώπη και που θα συμμετέχει στην επιστημιστική ισορροπία σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό σημαίνει και απαιτεί δεσμεύσει πολιτικέ ω προ τη ρύθμιση των αγορών, και αυτό είναι το θέμα που συζητούμε σήμερα. Δηλαδή, αν θα πρέπει και εμεί στι συζητήσει μα στο ευρωπαϊκό επίπεδο να ενσωματώσουμε αυτέ τι ιδέε και τη στιγμή που θέλουμε που γίνεται λόγος για κατάργηση αυτής της διάστασης της ε, παραγωγής τροφίμων στην Ευρώπη επανέρχεται η επικαιρότητα της ε, διατροφικής αλληλεγγύης και της προστασίας αυτών των 30 εκατομμυρίων Ευρωπαίων που υποσυτίζονται στην σημερινή εποχή. Μεγάλες λοιπόν κατευθύνσεις, πράσινη γεωργική πολιτική χάρη στην έκθεση που επεξεργαζόμαστε. Ναι, θα πρέπει να σωματωθεί η περιβαλλοντική πτυχή στο χώρο της γεωργίας και αυτό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μέσα από έναν πρώτο πυλώνα που ενσωματώνει το περιβάλλον ε, στις, ε, ε, στους όρους του και δεύτερον, και αυτό είναι προϊόν μακρών διαπραγματεύσεων, ένα, ένα αντικείμενο στο οποίο εγώ δεσμεύτηκα από την αρχή, ήταν η σταδιακή μείωση των ενισχύσεων και η ανακατανομή τους κατά τρόπον, ισοδύναμο, κατά τρόπον ισότιμο με ε, θεώρηση και της, ε, του παράγοντα απασχόληση, δηλαδή θα πρέπει να δείξουμε ότι μπορεί η γεωργία να συμβάλλει στην απασχόληση και της προσέγγισης ε, της παροχής δημόσιου αγαθού. Γιατί με, μόνο με αυτά τα δύο δεδομένα μπορούμε να φτάσουμε σε μια ουσιαστική ε, ε, απόφαση και αυτό το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια γιατί το πιστεύω ακράδαντα. Η έκθεση δε κατά λίγο ε, έχει αξία μόνο εάν ο προϋπολογισμός που έχει ε, οριστεί για την γεωργία μέχρι τώρα παραμείνει απαράλλαχτος και αν ισχύσουν τα όσα μας είπε ο κύριος Επίτροπος για το δεύτερο πυλώνα που θα πρέπει να περισταλεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Λεφόλ. Για δύο λεπτά ακόμη ο κύριος Λιού. Ο κύριος Λάιον, συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και συνεισηγητές και συνάδελφοι. Η έκθεση αυτή στην αρχική της μορφή νομίζω ο Ρόμπερτ Μπέρνς, ο εθνικός ε, ποιητής ε, της Σκοτίας θα την περιέγραφε ως ε, ένα τέρας μέσω των προσπαθειών του Άλμπερτ Ντες ε, τους τελευταίους μήνες έχουμε μία έκθεση με ουσία και πολλά στοιχεία που μπορούμε να στηρίξουμε. Θεωρούμε όμως πως υστερεί σε ένα σημαντικό τομέα. Δεν απαντά στο μιλιώδες ερώτημα που ρωτούν οι φορολογούμενοι και καταναλωτές που πληρώνουν την κοινή κυριολογική πολιτική. Ποια, ποιες είναι οι άμεσες αποσυνδεδεμένες πληρωμές τι χρειάζονται. Δεν υπάρχει πλέον σύνδεση με την παραγωγή καθώς έχει αποσυνδεθεί. Υπάρχει σύνδεση με, τα δημόσια αγαθά μέσω της πολλαπλής συμμόρφωσης, αλλά δεν απαντά αυτό στην ερώτηση και θεωρώ πως η έκθεση θα έπρεπε να έχει πάει λίγο πιο μακριά ως προς αυτό ακριβώς το ερώτημα με το να στηρίζει την ιδέα πιο στοχευμένων άμεσων ενισχύσεων που θα σχετίζονται με ένα πιο βιώσιμο και ανταγωνιστικό μοντέλο των άμεσων πληρωμών σε σύνδεση με τις ε, μειονεκτικές ε, περιοχές και το λεγόμενο πρασίνισμα της, της κοινή γεωργικής πολιτικής. Νομίζω πως αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα και να απαντήσουμε σε τι χρησιμεύουν οι άμεσε πληρωμές και έτσι ακυρώνει αυτά τα οποία ακούστηκαν για πλαφόν γιατί βεβαίως εάν γίνει αυτό σε όλες τις άμεσες ενισχύσεις τόσο όσο μεγαλύτερο είναι ο αγρότης τόσο περισσότερο και η ενίσχυση. Θεωρώ πως η έκθεση πάει προς αυτή την κατεύθυνση και καλωσορίζω αυτή την κίνηση θα έλεγα. Ελπίζω να μπορέσουμε να τη βελτιώσουμε αύριο και αν γίνει αυτό η ομάδα μας ευχαρίστως να τη στηρίξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λάιον. Ακολουθεί ο κύριος Νίκολσον επίσης για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δράτω με τις ευκαιρίες να συγχαρώ και τον εισηγητή. Απέδειξε στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ότι έχει πολύ ε, υπομονή γιατί πολλοί ε, προσπαθούσαν να το χτυπήσουν εκείνο το διάστημα και παρόλα αυτά ήταν πολύ αποφασιστικό στα καθήκοντά του και το κατέληξε στο αποτέλεσμα. Καταρχάς ε, χαίρομαι που θα υπάρχει μια δομή πυλώνα 2 γιατί νομίζω ότι σε αυτό συμφωνήσαμε όλοι. Άκουσα και τα όσα είπαμε για το πρασίνισμα και όταν αναφερόμαστε στο πρασίνισμα, ο καθένας ε, αντιλαμβάνεται διαφορετικά πράγματα στις διάφορες χώρες. Θα πρέπει κάπου να το σκεφτούμε όλοι. Δεν είναι απλώς ε, μία εύκολη ατάκα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να ε, τραβήξουμε την προσοχή, γιατί θα έχει πολύ σημαντικές συνέπειες για το μέλλον. Ο Λεφόλ έχει δίκιο. Ε, εάν δεν υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε και πολλά πράγματα σε αυτούς τους τομείς. Και ναι, πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι και πρέπει να επιδείξουμε υπευθυνότητα ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν θέλουμε να προχωρήσουμε στο νομοθετικό κείμενο που θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πόρο αργότερα και αυτό θα αποτελέσει τεράστια πρόκληση για μας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι για πρώτη φορά θα έχουμε ευθύνη και θα είμαστε τμήμα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Από αυτό το πρίσμα λοιπόν θα πρέπει να πω ότι εγώ είμαι αντίθετο στο παρόν κείμενο όταν αναφερόμαστε στα χάσματα. Θα υποστηρίξω τροπολογίες που ε, κατατέθησαν για να μειώσουμε το βαθμό αυτό. Ε, και όπω σα είπα, δεν θα υπάρξει κανένα όφελο αν δεν έχουμε και τον αντίστοιχο προπολογισμό. Θα πρέπει όμω να εξετάσουμε και πώ θα δαπανίσουμε τα κονδύλια. Θα δαπανούμε όσο το δυνατόν καλύτερα αυτή τη στιγμή. Μήπω πάνε πάρα πολλά σε διοικήσει, γραφειοκρατία. Μήπω ε, δεν δίνονται αρκετά στους ανθρώπους ε, που αναφέρονται και στην επιστημιστική ασφάλεια όπως και στο πρασίνημα. Τι κάνουμε για να βελτιώσουμε την επιστημιστική ασφάλεια. Μπορεί να υπάρξει κρίση τα επόμενα δέκα χρόνια. Έχουμε λιγότερους γεωργούς, λιγότερους ανθρώπους που ασχολούνται με τον ταμέα και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη για το μέλλον. Ευχαριστώ κύριε Νίκολσον. Για δύο λεπτά ο κύριος Χόισλινγκ. Ε, ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Κατά την απόψή μας η έκθεση πάει προς σωστή κατεύθυνση. Η ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική πρέπει να γίνει πιο δίκαια. Πιο... Δίκαιη, με συγχωρείτε. Να λάβει υπόψη το περιβάλλον και βεβαίως να λάβει υπόψη τους στόχους κλίματος και βιοπικιλότητας και αυτό νομίζω αναφέρεται στην έκθεση. Θα πρέπει λοιπόν να έχει περιβαλλοντικές επιδόσεις, τότε είναι διατεθειμένος ο φορολογούμενος να πληρώσει. Χρειαζόμαστε δικαιότερη κατανομή μεταξύ των εκμεταλλεύσεων και των κρατών μελών και αυτό νομίζω περιέχεται στην έκθεση. Δύσκολη διαδικασία, 1300 ε, τροπολογίες αλλά νομίζω πως έχουμε επιδείξει μεγάλη διάθεση συμβιβασμού. Νομίζω έχει δείξει το Κοινοβούλιο πως είναι ικανό να ασκήσει πολιτική εδώ πέρα. Κάποια πράγματα μπορούσαν να είναι σαφέστερα για εμάς. Παραδείγματο χάρη ποιοι είναι οι όροι σύμφωνα με τον πρώτο πυλώνα, προστασία των εδαφών κτλ. Εντάξει τώρα θα τα δει αυτά η Κομισιόν στην τελική διαμόρφωση. Επίσης ε, υπάρχει η φθήνουσα αναλογικότητα, καθώ πρέπει να κάνουν περισσότερα με λιγότερα λεφτά ή μεγαλύτερε εκμεταλλεύσει. Ενισχύεται ο ρόλο ε, των γεωργών και σημαντικό είναι το θέμα του ελλείμματο των λευκομάτων. με τα... των πρωτεϊνών. Βεβαίως σημαντικό είναι να δούμε τον ισχυρό δεύτερο πυλώνα αγροτική ανάπτυξη, περιβαλλοντικά ζητήματα και ενίσχυση των περιφερειών. Πράγματα που θέλει να περικόψει ο κ. Μπαρόζο. Εδώ πέρα θα αντισταθεί το Κοινοβούλιο. Εκεί πέρα ακριβώς βρίσκονται οι ευκαιρίες των μειονεκτικών περιοχών και της ε, αγροτικής ανάπτυξης. Ευχαριστούμε κύριε Χόισλινγκ. Ο κύριος Λέιερικ για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Η έκθεση που μας ε, κατατέθηκε περιγράφει τη νέα κυριγυρική πολιτική, προοδευτική διαμόρφωση των δημόσιων πιστώσεων για την απασχόληση και το περιβάλλον, αναγνώριση της δημόσιου, του χαρακτήρα δημόσιας υπηρεσίας προσφέρει η κοινωνική πολιτική, την παρουσία ω ενεργού φορέα και παράγοντα του γεωργού. Όμω έχουμε και παλιά κακή παράδοση ω προ τον εργαζόμενο στην γεωργία. Είναι μεγάλα τα δράματα που ζούμε ακόμη αυτή τη στιγμή στην Ήπεθρό μα και μπορεί να μην επαρκούν τα μέτρα αυτά. Πρέπει λοιπόν τότε να μπορούμε να επιστρέφουμε σε μηχανισμούς ενισχύσεων που θα εξασφαλίσουν ελάχιστες τιμές βάσης για το μικρό και μεσαίο παραγωγό. Η αποτελεσματικότητα, οι προκλήσεις οικολογικές σημαίνουν ότι θα πρέπει ταυτόχρονα να, να εγκαταλείψουμε την ε, άκρατη ελευθερία στην οικονομία της αγοράς, στο σύστημα των ελεύθερων ανταλλαγών που καταστρέφουν τις μικρές κυρίως εκμεταλλεύσεις και να επανέλθουμε σε ένα σύστημα διαφορετικό συνεργασίας που θα εισάγει ε, τέλη στην εισαγωγή των προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να επιμείνουμε... Κλείνει το μικρόφωνο του ομιλητή. Ευχαριστώ κύριε Λουιαγκ Το λόγο τώρα έχει... Η κυρία Μόρβα για ε, διαδικαστικό σας παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν μπορέσαμε να ακούσουμε την διερμηνία στα αγγλικά της τελευταίας παρέμβαση του κυρίου Λογιαρίκ. Και ήθελα να τον ακούσω. Μήπως θα μπορούσε, αν δεν ε, κουράζουμε πολύ τον ομιλητή, να ακούσουμε την ε, διερμηνία, αν μπορείτε να κάνετε μια χειρονομία κι εσείς από πλευρά σας. Ο Πρόεδρος, υπήρξε κανείς άλλος ο οποίος δεν άκουσε αγγλική διερμηνία. Μήπως ήταν τοπικό το φαινόμενο. Μήπως είναι μόνο η πίσω, τα πίσω έδρανα. Όχι. Προφανώς ε, ήταν μία σύγχυση σχετικά με τα κανάλια. Συνηθίζεται. Παρακαλώ, έχετε κατανόηση, αλλά υπάρχει web stream. Ε, άρα πιστεύω ότι η διερμηνία κάπου θα βρεθεί. Τώρα το λόγο έχει ο ε, κύριος Φοντάνα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητέ Επίτροπε. Ε, συγχαίρω τον εισηγητή, μαζί με τους κοιόδης εισηγητές, για τη δύσκολη δουλειά. Είμαστε ικανοποιημένοι που στο εσωτερικό της έκθεσης αυτής υπάρχουν αναφορές στις ε, ορεινές περιοχές, στις προβληματικές περιοχές. Ε, υπάρχει υποστήριξη για τις ε, μικρές επιχειρήσεις που είναι σημαντικό αυτό γιατί έχουν μεγάλη σημασία και για όλη μας την επικράτεια αλλά και για την ποιότητα των προϊόντων που παράγουν αυτές οι μικρές επιχειρήσεις. Επίσης μας ικανοποιεί το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές αναφορές στους νέους αγρότες, που είναι το μέλλον ουσιαστικά της γεωργίας. Όλοι ξέρουμε όμως ότι η μεγάλη μάχη θα δοθεί στον προπολογισμό. Ε, πίτροπε, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε η ΚΑΠ να έχει περικοπές στον προπολογισμό της, γιατί αυτό σημαίνει ότι η γεωργία δεν αξίζει πια τίποτα στην Ευρώπη. Και αν αξίζει λιγότερο στην Ευρώπη, σημαίνει ότι αξίζουν και τα γεωργικά προϊόντα λιγότερο στην Ευρώπη και άρα και όλη μας η διατροφή αξίζει λιγότερο. Νομίζω, κύριε Επίτροπε, ότι τώρα πρέπει να θέσουμε και ένα ερώτημα για τι εισαγωγέ που δεν εντάσσονται στην ΚΑΠ, αλλά είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο μαζί με την ΚΑΠ. Γιατί αν εισάγουμε ε, προϊόντα χαμηλή ποιότητα και χαμηλού κόστου, η δική μα γεωργία πρόκειται να αποτύχει. Ευχαριστώ κύριε Φοντάνα. Τώρα για μία λεπτά ο κύριος Τόντς. Η κυρία Τόντς, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ τον κύριο Ντές για αυτή την ε, πολύ καλή έκθεση και όπως και άλλοι ομιλητές ε, θα ήθελα να τονίσω τη σημασία ε, του καλού προπολογισμού για την μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική για να εξασφαλίσουμε τη διατροφική ασφάλεια διότι μέχρι το 2050 θα χρειαστούμε μία 50% αύξηση στην ε, ε, παραγωγή τροφίμων και στην Ευρώπη ε, δεν πρέπει να κάνουμε κάτι το οποίο ε, θα ε, βλάψει τη βάση παραγωγής την οποία έχουμε ήδη. Γι' αυτό και εγώ συμφωνώ με την δομή σε δύο πυλαώνες και την προσφορά στηρίξεως από τον Επίτροπο. Πρέπει όμως να σας πω ότι δεν θα ήθελα να υπάρξει μία επιβολή περισσότερων βαρών εις τους γεωργούς μας και γι' αυτό θα ήθελα να υπάρξει σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο μία ευελιξία η οποία να είναι προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ευχαριστώ. Κυρία Ντότς, το λόγο έχει τώρα για δύο λεπτά ο κύριος Λαβία. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η έντονη δουλειά που έκανε ο εισηγητής και οι σκιώδεις εισηγητές, ε, τους οποίους συγχαίρω, φτάνει στην τελική ευθεία σήμερα. Μία νέα ΚΑΠ ε, σημαίνει πάρα πολλά για την Ευρώπη, για το μέλλον της γεωργίας της, για την επιβίωση πολλών ε, εκτάσεων της υπαίθρου. Η νέα κοινή ε, πολιτική θα πρέπει να επιτρέπει στους Ευρωπαίους πολίτες να υποφελούνται από μια σωστή παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και για να υλοποιηθούν οι στόχοι θα πρέπει να υπάρξουν νέα μέσα, νέα εργαλεία, πιο αποτελεσματικά. Κυρίως πιο απλά για τους γεωργούς να έχουν πιο εύκολη πρόσβαση στους ε, πόρους και λιγότερο γραφειοκρατικό άχθος. Χρειαζόμαστε επίσης εργαλεία για την αγορά, για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις ε, επαναλαμβανόμενες δυστυχώς κρίσεις, ε, καθώς και εργαλεία πρόληψης των κινδύνων που είναι κλασικά στην, στο γεωργικό τομέα. Επίσης χρειαζόμαστε μια κάπη για τους νέους που εξασφαλίζουν τη γεωργία του μέλλοντος. Επιλέξαμε να προωθήσουμε την βιοπικιλότητα και την, τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων εδαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω μιας πολιτικής ανάπτυξης της υπαίθρου που μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε όλες τις φυσικές δυνατότητες αλλά και τους ανθρώπινους πόρους. Θα πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικές και ανταγωνιστικές να είναι οι εκμεταλλεύσεις μας οι γεωργικές. Γι' αυτό τονίζω στην Κομισιόν ότι θα πρέπει στην ανάπτυξη της υπαίθρου να έχουμε μέτρα για την μεταφορά τεχνολογίας με βάση τα όσα ψηφίστηκαν στην ε, Επιτροπή Γεωργίας, θέλω να τονίσω τη σημασία να εισαγάγουμε ε, μέγιστη, μέγιστα όρια α, στις άμεσες πληρωμές των μεγάλων επιχειρήσεων. Θα πρέπει να υπάρχει βαθμία μείωση των ενισχύσεων ανάλογα με το μέγεθος της ε, ε, επιχείρησης πάνω από ένα συγκεκριμένο κατόφλι. Ούτω ή άλλω οι μεγάλε αυτέ ε, οι, οι από μεγάλε οικονομίε κλίμακα. Θα πρέπει να υπάρχει επαρκή χρηματοδότηση τη κοινή ε, γεωργική πολιτική. Δεν μπορούμε να δεχτούμε εμεί ω Κοινοβούλιο τη μείωση των πόρων για την ανάπτυξη τη υπαίθρου. Ευχαριστώ. Ε, ο κύριο Λούχαν θέλει μπλε κάρτα. Mm -hmm. Θέλετε να απευθύνετε μια ερώτηση στον κύριο Λάβια. Κύριε συνάδελφε, Catch the Λοιπόν, ο επόμενος ομιλητής για ένα λεπτό, ο κύριος Κάπουλα Σάντος. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Οι σοσιαλιστές θέλουμε η κοινή γεωργική πολιτική είναι πιο δίκαιη. Ιδιαίτερα μάλιστα σήμερα όπου τα θέματα νομιμότητας σε σχέση με τη διατροφική ασφάλεια έχουν πάρει μια ιδιαίτερη σημασία. Καταφέραμε να συμπεριλάβουμε στην έκθεση τις κύριες ανησυχίες μας. Για παράδειγμα το πώς θα διατηρήσουμε μια κοινοτική κοινή γεωργική πολιτική η οποία θα πρικοδοτείται κατάλληλα. Υπογραμμίζω ότι για αυτό το θέμα δεν θα δεχτούμε να αφαιρεθούν πόροι από την κοινή γεωργική πολιτική. Θέλουμε να γίνεται καλύτερη κατανομή της στήριξης μεταξύ των χωρών μελών και των γεωργών και να υπάρξει ένα νέο σύστημα αποσύνδεσης που να σέβεται το περιβάλλον. Θέλουμε επίσης να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην απασχόληση και να προσανατολίσουμε την κοινή γεωργική πολιτική στους πραγματικούς αγρότες και στους μικρούς αγρότες. Είναι αλήθεια ότι με τον ενισχυμένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τώρα μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας θα καταφέρουμε να κάνουμε πράξη τους στόχους αυτούς που προς το παρόν είναι μόνο θεωρία. Το λόγο για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και στον κύριο Ντες για την τόσο καλή του δουλειά. Υπάρχει ένα σημείο που θέλω να αναφέρω σε σχέση με την κοινή γεωργική πολιτική. Και αυτό είναι οι μαζικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ολόκληρη η ανθρωπότητα. Περιβάλλον, βιοπικιλότητα, ευτροφισμός στο είδωρ, να μερικά θέματα που έχω να αναφέρω. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι οι γεωργοί εκείνοι οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, προστατεύοντας το περιβάλλον προκειμένου να μας βοηθήσουν να επιβιώσουμε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να βρούμε τους καλύτερους δυνατών μηχανισμούς. Η χρήση λοιπόν των περιβαλλοντικών μέσων που χρησιμοποιούν οι γεωργοί και για τους οποίους πρέπει να πληρώσουν οι γεωργοί είναι αυτό που θα μας βοηθήσει. Αλλά επειδή ακριβώ πρέπει να επενδύσουν σε αυτούς οι γεωργοί, θα ήθελα στο μέλλον και εμείς να αλλάξουμε λιγάκι τακτική και αντί να επιδοτούμε το εισόδημα, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξηγήσει κανείς σήμερα, να φροντίσουμε να πληρώνουμε την πραγματική δουλειά που κάνουν οι αγρότες. Να περάσουμε δηλαδή από την επιδότηση στην πληρωμή πραγματικών υπηρεσιών. Προφανώς δουλειά της γεωργίας και των γεωργών είναι να παράγουν τρόφιμα. Τρόφιμα, αρκετά τρόφιμα, καλή ποιότητας τρόφιμα. Πιστεύω ότι τα τρόφιμα πληρώνονται στην αγορά. Η προστασία του περιβάλλοντος όμως δεν πληρώνεται από την αγορά. Τώρα για ένα λεπτό ο κύριος Φορτσιοκόφσκι θα πάρει το λόγο. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η έκθεση του κυρίου Ντες ε, από πολλές πτυχές είναι πάρα πολύ καλή, αλλά υπάρχει και μια άσχημη πτυχή γιατί αρνείται την ιδέα της δίκαιης ε, εξισορρόπησης των άμεσων πληρωμών. Με αυτόν τον τρόπο οι φτωχοί παίρνουν μεγαλύτερη βοήθεια από τους ε, φτωχούς. Η γεωργία στα νέα κράτη-μέλη γίνεται όλο και πιο αδύναμη και μεγάλα κομμάτια γης δεν χρησιμοποιείται στην Πολωνία, Λιθουανία, Σλοβακία και αλλού. Γι' αυτό κάνω έκκληση στους συναδέλφους από τα παλιά κράτη-μέλη να σταματήσουμε αυτή τη διάκριση, να πληρώσουμε το ίδιο, τις ίδιες άμεσες δηλαδή πληρωμές, ε, σε όλα τα νέα κράτη-μέλη. Στρέφομαι στους συναδέλφους από τη Γαλλία. Θέλετε, θέλατε εσείς ελευθερία, αδερφοσύνη και, ελε... και χωρίς όμως ισότητα δεν υπάρχει αδερφοσύνη. Αμέσως απαντάει η Γαλλία. Δύο λεπτά κύριε Εμποβέ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί φίλοι, ναι, σύμφωνο ώστε με την ε, αδελφοσύνη και ε, την ε, συναδελφικότητα να υπάρξει και ισότητα με τα νέα μέλη από την Ανατολική Ευρώπη. Προχωρήσαμε πολύ με την έκθεση αυτή. Υπήρχε μία αντιπαράθεση στην αρχή αλλά φτάσαμε σε μία συμφωνία και η συμφωνία αυτή επιτρέπει να προστατεύσουμε το συνολικό πρόγραμμα και αυτό είναι το προτέρημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το επιτύχαμε, δεν ήταν εύκολο και ευχαριστώ τον εισηγητή κύριο Ντέ και τους βουλευτές. Σε αυτό το κείμενο τονίζουμε την ανάγκη να υπάρξει ισότητα, δικαιοσύνη και ισοτιμία μεταξύ των ε, παραγωγών και των περιοχών. Το διακηρύξαμε και είναι βασικό και να μπορέσουν να αναπτυχθούν τα μικρά αγροκτήματα που είναι απαραίτητα για την ποιότητα και την βιοπικιλότητα των ε, διαφόρων περιοχών ήταν πολύ βασικό. Επίσης πρέπει να έχουμε αγρονομική ε, γεωργία είναι εγγεγραμμένο στα διάφορα κείμενα πρέπει τώρα να εφαρμοστεί για να μπορέσει να υπάρξει εφικτή και βιώσιμη γεωργία για τις επόμενες γενιές. Αυτό που μας ανησυχεί σήμερα είναι ότι υπάρχουν απειλές για τον προϋπολογισμό πρέπει να απαντήσουμε σαφώς και περιμένουμε να προχωρήσουμε στη δεύτερη φάση δηλαδή να υπάρξει η ε, νομοθετική συζήτηση διότι σε αυτή τη συζήτηση όντως θα δούμε προς τα που κατευθυνόμαστε και αυτό περιμένουμε τώρα. Θέλω να τελειώσω και ε, να ε, εκφράσω το θυμό μου έναντι της θέσεως της ε, Γερμανίας διότι μειώσαμε δια του 5 το, τη βοήθεια στους στοχότερους στην Ευρώπη. Πρέπει να βοηθήσουμε τα 80 εκατομμύρια Ευρωπαίους που δεν τρώνε όσο χρειάζονται χρειάζονται. Σας παρακαλώ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Για ένα λεπτό ο κύριος Ρούμπιξ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μια μεγάλη προσπάθεια έχει γίνει. Α, όμως η έκθεση που παρουσιάσαμε είναι πολύ γενικόλογη. Εστιάζει σε μια νέα κατεύθυνση στη γεωργία, της πράσινης γεωργίας. Αυτό θα μπορούσε να είναι ε, ένα σωσίβιο για τους παραγωγούς που δεν παράγουν ουσιαστικά για να έχουν κάποιο εισόδημα. Κατά τη γνώμη μου, όταν αυτή η έκθεση εφαρμοστεί, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε κάποια ζητήματα, την ποιότητα των τροφίμων, την επιδείνωση της κατάστασης της ε, γης. Επίσης ε, δεν υπάρχουν ε, ορισμοί για τις άμεσες πληρωμές, για, τους οικογενειακούς, για τις οικογένειες που δουλεύουν στη Γεωργία, για τους νέους γεωργούς. Δηλαδή, δυστυχώς πολλοί γεωργοί δεν θα μπορέσουν να βρουν ερωτήσεις στα απαντήματα, στις, απαντήσεις ερωτήσεις του. Συγγνώμη. Ένα λεπτό παρακαλώ. Whilst the term greening of pillar 1 το πρασίνισμα του πρόσου πυλώνα μπορεί να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα σε ορισμένους αγρότες. Η πολιτική αυτή, αν είχε εφαρμοστεί φέτος, θα είχε καταλήξει μεγάλη καταστροφή για τις οδιές. Τα μέτρα αυτά δεν μπορούν να εφαρμοστούν καλά. Για να εφαρμοστούν καλά πρέπει να υπάρξει και αυστηρός έλεγχος, πράγμα που σημαίνει ότι τελικά αυτό που θα κάνουν οι αγρότες είναι να μοιραστούν τη δουλειά με τις συζύγους τους. Εξάλλου, οι αποταμιεύσεις δεν θα πάνε στα κράτη-μέλη που θα έχουν φροντίσει για τις αποταμιεύσεις αυτές. Η πρόταση ότι η πληρωμή αυτή θα φτάσει στους αγρότες που τους δικαιούνται δεν είναι αλήθεια. Δεν θα έχουμε αρκετά τρόφιμα. Αντίθετα, πρέπει να ενισχύσουμε και να βοηθήσουμε τους αγρότες να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες. Οι Μάλλον οι, ναι, οι σκληροί χειμώνε πρέπει να μα έχουν πείσει ότι δεν κινδυνεύουμε από τη θέρμανση του πλανήτη. Έχει το λόγο για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ αγαπητοί κύριοι ευρωβουλευτέ, Ορισ μένει θα είχαν διαφορετική άποψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση περί της ε, ενώσεως αυτής ε, διότι ε, τα, οι φόροι οι οποίοι καταβάλουν θα ήθελαν να διατίθενται μόνο για δημόσιους στόχους και μόνο προς δημόσιο όφελος. μαζί με ε, τις ε, ενισχύσεις της κοινή γεωργικής πολιτικής ε, το θέμα αυτό πραγματεύεται η έκθεση του κυρίου Ντες την οποία θα ψηφίσουμε αύριο. Ε, σχετικά με την ενίσχυση και τη στήριξη η οποία προβλέπεται ε, ανά επιφάνεια εκτάσεων και θα ήθελα να ε, σκεφτείτε ότι πρέπει να είστε δίκαιοι έναντι των πολιτών πρέπει να δεχθούμε το ανώτατο επίπεδο το πλαφόν πρέπει να το δεχτούμε και δεν πρέπει να στηρίξουμε τους κόκκινους και πράσινους βαρώνους Ευρωπαϊκής Ενώσεως Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η σημερινή συζήτηση έχει να κάνει με την πολύ σοβαρή αυτή έκθεση για την κοινή γεωργική πολιτική. Εγώ θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο το οποίο μας επηρεάζει και μπορεί να επηρεάσει και την ε, βιωσιμότητα των μέτρων που στηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής. Την επόμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει την πρότασή τη για τις δημοσιονομικές προοπτικές τη επόμενη για την περίοδο 2014. Αν ε, είναι σωστές οι πληροφορίες μου, Πρόθεση είναι να προτείνουν μείωση του γεωργικού κοινοτικού προπολογισμού. Γι' αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη μα ότι η έκθεση που θα εγκρίνουμε αύριο και με την οποία ζητάμε ακριβώ να διατηρήσουμε τι δαπάνε για την κοινή γεωργική πολιτική δεν θα ληφθεί υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ δεν βλέπω πώ είναι δυνατόν με ένα προπολογισμό ακόμα πιο περιορισμένο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλε τι προκλήσει που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό. Πώ είναι δυνατόν να είναι πιο πράσινη η γεωργία μα, πώ είναι δυνατόν να πετύχουμε του στόχου που θέλουμε με την προστιθέμενη αξία των δικών μα γεωργικών και εκνοτροφικών προϊόντων. Δεν βλέπω πώ θα γίνει αυτό. Δεν βλέπω πώ είναι δυνατόν με μια περιορισμένη ΚΑΠ να περιμένουμε, για να δώσω άλλο ε, παράδειγμα, να σταθεροποιήσουμε τι τιμέ. Χρειαζόμαστε μια γραμμή στον προπολογισμό η οποία να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει κρίσει που κάθε τόσο αντιμετωπίζουμε η ΚΑΠ πρέπει να πρικοδοτείται παρκώς, γιατί πέρα από τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που μας προσφέρει, σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι σαφές ότι ένα ευρώ, ένα ευρώ που επενδύεται στη γεωργία δημιουργεί 10 ευρώ πλούτο στον ε, τομέα των αγροτροφίμων. Γι' αυτό πρέπει να το λάβουμε πάρα πολύ καλά υπόψη μας αυτό όταν θα ετοιμάσουμε το νέο δημοσιονομικό μας πλαίσιο. Επιπλέον, χωρίς να ξεχνάμε ότι οι διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου απειλούνται. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε να έχουμε την παραγωγή που θέλουμε στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ο Δεκάστρο θα πάρει το λόγο για ένα λεπτό παρακαλώ. Κύριε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, με την έκθεση DES ξεκινάει μια νέα φάση στην ε, διαδικασία μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Μια έντονη προσπάθεια της Επιτροπής Γεωργίας που κράτησε πολλούς μήνες και για την οποία θέλω να ευχαριστήσω τον Άλμπερντες και όλες τις ε, κοινοβουλευτικές ομάδες για τη δουλειά του. Σήμερα το Κοινοβούλιο μπορεί να εκφράσει μια ξεκάθαρη φωνή για το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής. Μια κάπα στεναρή, απλή, ευέλικτη, πιο πράσινη, που συμπεριλαμβάνει και τους νέους ε, και την εργασία. Γι' αυτό ε, το λόγο, Επίτροπε, Μα ανησυχεί η μείωση του προπολογισμού του δεύτερου πυλώνα, κάτι που διαβάζουμε σε εφημερίδε. Αυτό είναι ασύμβατο και με το περιεχόμενο τη έκθεση ΔΕΣ και με την έκθεση για τι δημοσιονομικέ προοπτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση του κ. Γκαρίγκα, που ψηφίσαμε στην Ολομέλεια τι περασμένε εβδομάδε και που εισήγαγε για την κοινή γεωργική πολιτική την ε, σημαντική αρχή τη διατήρηση ε, του, σημαν... του σημερινού ποσού ε, πιστώσεων για την επόμενη περίοδο. Γι' αυτό θα ήθελα να μας ξεκαθαρίσετε τι είναι όλα αυτά τα νέα που ακούμε και αν εσείς έχετε διαφορετικό προσανατολισμό σε σχέση με αυτά που μας είπατε μέχρι σήμερα. για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι, ευχαριστώ τον εισηγητή για την καλή εργασία την οποία ναι έκανε και όσον αφορά το μέλλον της γεωργικής πολιτικής μετά το 2013 πρέπει να αποφασίσουμε πού θέλουμε να κατευθυνθούμε. Θέλουμε μια γεωργία η οποία θα είναι και οτόμα σύγχρονη, ε, υπεύθυνη και ε, θα λειτουργεί αποφασιστικά ή θέλουμε μια γεωργία η οποία θα είναι πάντοτε οπισθοδρομική και θα συνεχίσει έτσι. Γι' αυτό θα πρέπει για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα του μέλλοντος αντί να έχουμε ε, συνεχείς συζητήσεις ιδεολογικές να εφαρμόσουμε τεχνολογικές μεθόδους για να μην αλλάζουμε κατεύθυνση κάθε λίγα χρόνια αυτό επηρεάζει και επιδεινώνει την ε, οικονομική μας κατάσταση και οδηγεί σε νέα νομοθετικά μέτρα που χρειάζονται νέες επενδύσεις Χωρί χωρίς να αυξάνονται τα έσοδα. Δεν θα έπρεπε να μας ε, ενδιαφέρει αν μια επιχείρηση είναι μεγάλη ή μικρή, αλλά αν είναι υγιής και δουλεύει σωστά. Ε, αν λειτουργεί οικολογικά, αν μπορεί να χρησιμοποιεί σωστά τους σπόρους της. Δεν έχει σημασία πόσα ζώα υπάρχουν, αρκεί τα ζώα να είναι υγιή. Θα πρέπει να έχουμε επαρκή τρόφιμα καλής ποιότητα και σε καλές τιμές στο μέλλον στην Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη δεν είναι μόνη της στον κόσμο. Ο κύριος ε, μόνο για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Μπορούμε πια να δούμε ότι τι γίνεται όταν οι νέες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζουν την κοινή γεωργική πολιτική και δεν θα υπάρχουν πια διακρίσεις σε βάρος των χωρών αυτών. Ελπίζω να μην υπάρχουν στο μέλλον επιπλέον διακρίσεις. Δυστυχώς όμως βλέπω διακρίσεις ακόμα στην έκθεση του κυρίου Ντες. Βλέπω στήριξη για μια οροφή άμεσων πληρωμών, κάτι το οποίο αποτελεί διάκριση σε βάρος χωρών όπως είναι η Τσεχία, όπου έχουμε μεγάλες ε, ε καλλιέργειες, μεγάλες μονάδες εκτροφής. Είναι ένα μέτρο αυτό λοιπόν το οποίο κατά τη γνώμη μου θα μειώσει την αποτελεσματικότητα της γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η γεωργία πρέπει να παράγει τρόφιμα. Τώρα όμως τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι πολλοί πολιτικοί, ιδιαίτερα μεταξύ των ε, πρασίνων, που θέλουν οι γεωργοί να παράγουν βιοκαύσιμα. 1,5 λεπτό παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, συμφωνώ με τις ε, απόψεις των συναδέλφων και συγχαίρω τον εισηγητή. Η δουλειά του δεν ήταν εύκολη, ούτε για, ήταν εύκολη για οποιοδήποτε από εμά. Ε, πρέπει να θαυμάσω πολλά στοιχεία στην έκθεση αυτή, ιδίως όσον αφορά την συνέχιση των αμέσων πληρωμών στο σημείο 15, καλύτερη και δικαιότερη κατανομή μεταξύ κρατών και εντός των κρατών στην παράγραφο 16 και ερχόμενος από τη ε, Σκοτία είμαι ικανοποιημένος ε, για τη μνήα ε, στην παράγραφο 22 για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές και την, το, το θέμα της πολλαπλούς συμμόρφωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 44. Πολλά υπάρχουν να επικροτούμε στην έκθεση αυτή αλλά εάν αν ε, δεν υπάρξει η παράγραφος 1 δεν θα έχει νόημα όλο το υπόλοιπο κείμενο. Δηλαδή να υπάρχει φόρος ε, πολιτική με ικανοποιητικό προϋπολογισμό και ε, από ό,τι ξέρω ο πρόεδρος Μπαρόζο θέλει να περικόψει τους πόρους και θα χρειαστείτε όλους, κύριε Επίτροπε όλους τους συμμάχους στην Επιτροπή για να είμαστε φιλόδοξοι υπέρ των πολιτών. Η γεωργία της Ευρώπης είναι περίφημη και δεν πρέπει τώρα να την εγκαταλείψουμε. Ευχαριστώ. θα λόγο. Ευχαριστώ. Χαίρομαι για την έκθεση ΔΕΣ και για τόσα λέει για την μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Ψηφίζοντας την έκθεση αυτή δείχνουμε τι περιμένει από τις νομοθετικές προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ζωτική σημασία αν θέλουμε να έχουμε ικανοποιητική χρηματοδότηση της γεωργίας στο μέλλον. Πρέπει να έχουμε μία βιώσιμη κοινή γεωργική πολιτική, η οποία να βασίζεται σε δύο πυλώνες, ε, που θα βοηθήσουν τους αγρότες να παραμείνουν στη γη από τη μια και από την άλλη θα υπάρχει προστασία του περιβάλλοντος. Συγχρόνως θα αναπτύξουμε παρετέρω την οικονομία ε, στην Ήπεθρο και θα βοηθήσουμε και την τροφική αλυσίδα. Χρειαζόμαστε μέτρα για το πρασίνισμα της γεωργίας. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο και να υπάρχει καλός σχεδιασμός και ικανοποιητικός τρόπος αξιολόγησης αυτού του πρασινίσματος. Όλα αυτά πρέπει να τα τονίσουμε. Παρακαλώ. Κύριο Σκότα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Η κοινή γεωργική πολιτική είναι η ευρωπαϊκή πολιτική που περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χρειάστηκε να αλλάξει, να ανανεωθεί τα τελευταία χρόνια για να αντιμετωπίσει τις νέες οικονομικές συνθήκες και τις διεθνείς. Ε, αυτό έγινε χωρίς να ξεχνάμε ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε το εισόδημα των γεωργών και να αντιμετωπίσουμε τη συνεχή μείωση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Ε, μην ξεχνάμε από την άλλη ότι θέλουμε να εξασφαλίσουμε και την ποιότητα ε, των υδατινοπόρων, του περιβάλλοντο και των προϊόντων. Η μεταρρύθμιση που θα ψηφίσουμε αύριο είναι σημαντική για να συνεχίσουμε να ε, υποστηρίζουμε το εισόδημα των ε, αγροτών, όπω είπαν και οι συνάδελφοι. Όμω ο στόχο δεν είναι να μειώσουμε την άμεση ενίσχυση, αλλά να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στην παραγωγή και στην ύπεθρο, ούτω ώστε το σύστημα να είναι δίκαιο χωρί να αμφισβητούνται οι κανόνε του ανταγωνισμού. Σε ό,τι αφορά του στόχου τη ΚΑΠ στα πλαίσια τη ε, Στρατηγική Ευρώπη 2020, η ΚΑΠ μπορεί να συνεισφέρει ε, στη δημιουργία μιας ε, οικονομίας βιώσιμης, αντιμετωπίζοντας τις νέες προκλήσεις και λαμβάνοντας υπόψη τη ιδιαιτερότητα των 27 κρατών μελών. Για λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ανάγκη μιας ισχυρής ΚΑΠ είναι προφανής ο γεωργικός τομέας έχει σαφή προστιθέμενη αξία στην ευρωπαϊκή οικονομία. Διαδραματίζει πολυλειτουργικό ρόλο συμβάλλοντα στην παραγωγή δημοσίων αγαθών υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ θα πρέπει τουλάχιστον να παραμείνει στα ισχύοντα επίπεδα και να διασφαλιστεί η αντιστοιχεία πόρων και στόχων της νέας ΚΑΠ. Η κατανομή των πόρων της ΚΑΠ μεταξύ των γεωργών στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία καταλαμβάνει κυρίαρχη θέση στο δημόσιο διάλογο χρήζει προσοχής. επ' αυτού απορρίπτεται ευρέως ο καθορισμός ομοιομόρφου ύψους ενισχύσεως σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης το λεγόμενο flat rate. απαιτούνται κατά τη γνώμη μου αντικειμενικά κριτήρια ώστε να ληφθούν δεόντως υπόψη ιδιαιτερότητες του γεωργικού τομέα στα επιμέρους κράτη μέλη της ένωσης. επίσης θετικές είναι οι προτάσεις για θέσπιση οροφής στο ύψος των αμέσων πληρωμών, καταβολή ειδική ενίσχυσης στους μικρούς γεωργούς και καταβολή ενισχύσεων μόνο στους ενεργούς γεωργούς. Τα μέτρα οικολογικής πλαισίωσης θα πρέπει να είναι απλά στην εφαρμογή τους, να συνοδεύονται από επαρκές αντιστάθμισμα και να μην δημιουργούν επιπρόσθετο διοικητικό άχθος. Η εντυνόμενη αστάθεια των γεωργικών αγορών καθώς και η κλιματική κίνδυνη και οι διατροφικές κρίσεις επιβάλλουν την ενεργοποίηση αποτελεσματικών εργαλείων. Τα ισχύοντα μέτρα αγοράς θα πρέπει να ενισχυθούν. Επίσης χρειάζεται ένα μόνιμο ταμείο διαχείρισης κρίσεων. Θετική είναι η πρόταση για το νέο εργαλείο σταθεροποίησης γεωργικού εισοδήματος. Τέλος, υπογραμμίζω την ανάγκη αποτελεσματικών μέτρων υπέρ των νέων γεωργών. Ευχαριστίες στον εισηγητή, στον Άλμπερτ για το δύσκολο, συνθετικό έργο που επιτέλεσε και κύριε Επίτροπε, αποδυνάμωση της ΚΑΠ θα προσκρούσει στην πολιτική εναντίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω αυτό είναι το διακομματικό μήνυμα του σώματος και αυτό πρέπει να ληφθεί πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Παπαστάμκο. Η κυρία Ρόντους, για ένα λεπτό παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ τον εισηγητή και χαίρομαι διότι μια σοσιαλιστική ε, υπογραφή ε, διαφαίνεται στην έκθεση αυτή. Θέλουμε μια οικολογική ε, γεωργική πολιτική, θέλουμε πρασίνισμα και την θέλουμε στον πρώτο πυλώνα. Διότι δεν φτάνει το ισχύον σύστημα για να μπορέσει να γίνει αποδεκτό από κοινωνία αλλά είναι κάτι το οποίο χρειαζόμαστε. Ο ύψιστος στόχος μας πρέπει να έχουμε μια βιώσιμη παραγωγή τροφίμων στην Ευρώπη και έναν ενεργό χώρο της υπαίθρου και της γεωργίας. Ε, χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται στη γεωργία και θα την πονέσουν διότι υπάρχουν ψήθυροι για σημαντικές μειώσεις των πόρων μέτρων της αναπτύξεως της υπέρθρου και αυτό είναι απαράδεκτο και στο μέλλον πρέπει να επιμείνουμε σε έναν ισχυρό δεύτερο πιόλωνα για τη γεωργία και όλα τα μέτρα δεν μπορούν να μειωθούν διότι τότε δεν θα υπάρξει μεταρρύθμιση, θα μείνουν όλα αυτά τα έχουν και αυτό είναι απαράδεκτο για τους πολίτες της Ευρώπης χρόνο, κυρία συνάδελφε. Ε, Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, δεν θέλω να σα διακόπτω, αλλά προσπαθήστε κι εσεί να σεβαστείτε το, την ροή, ε, τη χρονική σα παρακαλώ, τη συζήτηση. Ε, τώρα για ένα λεπτό, ελπίζω να είναι ένα λεπτό, ο, ο κύριο Έσχορφ έχει το λόγο. Thank you, President. Uh, President Ευχαριστώ. Το Κοινοβούλιο ζητάει να διατηρηθεί και να αυξηθεί ο προπολογισμό για τη Γεωργία. Αυτό είναι πολύ φιλόδοξο. Η καιρή είναι σκληρή και τα χρήματα δεν είναι άπειρα. Κατά τη γνώμη μου χρειάζεται περισσότερος ρεαλισμός όταν αποφασίζουμε για τον προπολογισμό του χρόνου. Πρέπει να επανέλθουμε στις πραγματικές προτεραιότητες της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ασφάλεια τροφίμων, βιοποικιλότητα, αλλαγές στο κλίμα, νέες τεχνολογίες και δημιουργία ενός κλάδου τροφίμων με ασφάλεια για όλους. Νομίζω ότι έχουμε χάσει την πορεία αυτή στην οποία προσπαθούσαμε να βρεθούμε με τις δύο προηγούμενες μεταρρυθμίσεις. Όμως χαίρομαι που μπορώ να πω ότι με τις προστάσεις του ο Άλμπερτ Ντες θέτει ένα πολύ λογικό πλαίσιο ε, πάνω στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε για επόμενες εκθέσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Τώρα για δύο λεπτά η κυρία Κέστιγκερ θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, στην έκθεση του Albert Dess προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη ε, του κλίματος στην ε, γεωργία και υπάρχουν ικανοποιητικές διαπραγματεύσεις που έγιναν στα θέματα αυτά και ελπίζω ότι θα γίνουν αποδεκτό και το ανώτατο επίπεδο και ελπίζω ότι δεν θα πρέπει όσοι δεν αιτιολογούν τους πόρους να τους λαμβάνουν Πρέπει να καταργήσουμε την γραφειοκρατία, να αναμορφώσουμε τα συστήματα και με αυτόν τον τρόπο να μπορούμε να προωθήσουμε σωστά τον τομέα μας διότι ε, ε, πρέπει να ε, αποδεχθούμε ότι οι καταναλωτές ζητούν να υπάρξει βιωσιμότητα στον τομέα της γεωργίας και γι' αυτό πρέπει να υπάρξουν επαρκή οικονομική πόλη. Γι' αυτό και θα αντιταχθώ σε οποιαδήποτε μείωση του προϋπολογισμού. Ε, εάν ε, ο κύριος Μπαρόζο πάρει το κόκκινο μολύβι να διαγράψει τις, ε, τους πόρους της γεωργίας τότε θα του κόψει το νήμα της ζωής της γεωργίας και αυτά ήδη έχουν επηρεάσει τον σχετικό πυλώνα γι' αυτό και θα πρέπει το, ο πρόεδρος να ακούσει τη φωνή αυτού του Ευρωκοινοβουλίου Κοινοβουλίου και να παραμείνει η πολιτική αυτή κοινοτική διότι όσο υπάρχει αυξανόμενος ανταγωνισμός δεν μπορούμε να μειώνουμε τους πόρους ε, και να ζητούμε περισσότερα από τους γεωργούς μας. Το αντίθετο πρέπει να γίνει. Στον δεύτερο πυλώνα πρέπει να προωθήσουμε την καινοτομία και αυτό θα βοηθήσει τον τομέα της υπαίθρου. Θα πρέπει η οι νέοι ε, γεωργοί να μπορέσουν επίσης να δραστηριοποιηθούν για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν το μέλλον της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Γκαρσία Πέρες έχει το λόγο για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή συζήτηση δείχνει ότι το σώμα μας στηρίζει μια ισχυρή και κοινοτική κοινή γεωργική πολιτική που να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της διατροφικής ασφάλειας, του περιβάλλοντος και της απασχόλησης στην Ήπεθρο. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας, και νομίζω ότι αυτό θα κάνει και το σώμα, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε μειώσεις στον σημερινό προπολογισμό της ΚΑΠ. Χρειαζόμαστε μια επαρκή οικονομική χρηματοδότηση για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτές. Πρέπει να είμαστε σε θέση να εξασφαλίσουμε εισόδημα στους αγρότες μας και να διασφαλίσουμε μια αγορά η οποία να έχει σταθερές τιμές. Βέβαια δεν μπορώ να ξεχάσω και αυτά τα οποία έγιναν τις τελευταίες εβδομάδες στον τομέα των οποροκυπευτικών Πράγμα που σημαίνει ότι η καινούργια ΚΑΠ πρέπει να διαθέτει μέσα για να ανταποκρίνεται σε κρίσει που μπορεί να πλήξουν οποιοδήποτε τομέα τη. Μέσα τα οποία να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τι ανάγκε του κλάδου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα το λόγο για ένα λεπτό η κυρία Γκίρλινγκ θα πάρει το... Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Ντές για την πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ διαφωτιστική έκθεση. Ε, προφανώς ε, για... Ε, σε ένα τόσο περίπλοκο θέμα υπάρχουν ζητήματα με τα οποία συμφωνούμε ε, και ζητήματα με τα οποία συμφωνούμε. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει απόλυτη λογοδοσία όταν ξοδεύουμε το 42% του κοινωνικού προπολογισμού τη γεωργία. Αυξάνονται πολύ έντονα μερικέ φορέ οι τιμέ των τροφίμων και υπάρχουν προβλήματα στην προμήθεια. Ε, γι' αυτό εμείς θέλουμε μια ΚΑΠ η οποία θα εστιάζει στην αυξημένη παραγωγικότητα και στην αποτελεσματικότητα. Ναι, θα πρέπει να ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον. Εγώ είμαι μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και το ξέρω. Αλλά υπάρχει κίνδυνος να δημιουργήσουμε μια έκθεση που είναι πολύ ρητορική. Μιλάμε για το πρασίνισμα, ας πούμε, το, του πυλώνα 1. Μιλάμε για πράγματα τα οποία ξεχνάνε την ε, πραγματική εστίαση. Δεν θέλω να πληρώνουμε τις μεγάλες ε, εκμεταλλεύσεις. Ε, με αυτόν τον τρόπο θα θεσμοθετήσουμε την αποτελεσματικότητα και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για κάτι τέτοιο. για δύο λεπτά παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι. Καταρχήν ε, και αυτό το κάνατε όλοι ε, πρέπει να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή για την προσήλωση που ε, αφιέρωσε σε αυτή την έκθεση κατά τρόπον ώστε να καταλήξει σε αυτούς τους συμβιβασμούς. Δεν ήταν κάτι εύκολο αλλά έχουμε καλούς συμβιβασμούς τώρα. Είμαστε υπέρ μιας βιώσιμης και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής γεωργίας δηλαδή να παράγουμε τρόφιμα υψής της ποιότητος αλλά συγχρόνως να παράγουμε ε, ε, ε, έναν χώρο ποιοτικό, πολιτιστικό που θα αναζωογονεί και θα βοηθά όχι μόνο τη γεωργία αλλά και τον τουρισμό και άλλους τομείς. Και αυτή είναι μία παροχή την οποία προσφέρει η γεωργία σε ολόκληρη την κοινωνία αλλά η οποία δεν λαμβάνεται υπόψη επαρκώς από την κοινωνία. Είναι μια ξεχασμένη παροχή και αυτό οδήγησε στο ότι ο γεωργικός προϋπολογισμός πρέπει με κάθε τρόπο να μην μειωθεί περαιτέρω διότι χρειαζόμαστε περισσότερο πράσινο εις τον πρώτο πυλώνα αλλά δεν είναι δυνατόν αυτό να οδηγήσει για τις χώρες οι οποίες έχουν φιλόδοξα προγράμματα στο δεύτερο πυλώνα να ε, τιμωρηθούν και να υπάρχει βάρος τους διάκριση ε, γι' αυτό το λόγο. Θα πρέπει να είμαστε δίκαιοι προς όλους και όσον αφορά τα προγράμματα τα περιβαλλοντολογικά είναι δαπανηρά και αν διαβάσω τις εφημερίδες και αυτό το έθιξαν πολλοί συνάδελφοι είπαν ότι ο δεύτερος πυλώνας πρέπει να μειωθεί αλλά το απορρίπτω ναι μεν χρειαζόμαστε έναν ισχυρό πρώτο πυλώνα αλλά και έναν ισχυρό δεύτερο πυλώνα και στις προσπάθειες αυτές κύριε Επίτροπε θα σας βοηθήσουμε και θα σας στηρίξουμε. Κύριε Σταμπάτσι, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Τσόλο, κύριοι συνάδελφοι, η Κομισιό και το Συμβούλιο ε, λένε ότι θα πρέπει να υπάρχει επαρκής ε, επίπεδο χρηματοδότησης και εμείς θέλουμε μια επαρκή χρηματοδότηση για να στηρίξουμε και την πολιτική ανάπτυξη της υπαίθρου. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα και να υπάρχει συνειδητοποίηση για το περιβάλλον. Θα πρέπει να προωθήσουμε την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη. Όλα αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την κλιματική αλλαγή, να διαφυλάξουμε τη βιοπικιλότητα και να διαφυλάξουμε τους υδάτινου πόρους. Τα κράτη-μέλη στο μέλλον θα πρέπει να λάβουν περισσότερους πόρου για να ανακτήσουν την καθυστέρηση που έχουν, ειδικά σε τεχνολογικό επίπεδο, κυρίως μετά το 2013. Επίσης, τα νέα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τι ίδιε δυνατότητε και μετά το 2013. Δεν θα πρέπει επίση να ξεχάσουμε του μικρού παραγωγού. Ευχαριστώ πολύ Αποφύγαμε το χειρότερο, αλλά είχαμε 1267 τροπολογίες. Γι' αυτό και οι σοσιαλιστές προτίμησαν να καταθέσουν ένα ελάχιστο τροπολογιών και χαιρόμαστε που καταλήξαμε σε μια ισχυρή θέση μαζί με τον σκιώδη μα εισηγητή Στεφάν Λεφόλ. Μαζί με άλλε ομάδες λοιπόν και τον εισηγητή καταλήξαμε σε ένα φιλόδοξο συμβιβασμό. Αυτό που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό είναι η βοήθεια να πάει στους ενεργούς ε, ε, γεωργούς και όχι στους ιδιοκτήτε, ε, στους γεωκτήμονες δηλαδή, προκειμένου να προστατεύσουμε καλύτερα το περιβάλλον, να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τις υγιές και να αποφύγουμε παρατέρω κλιματικές αλλαγές. Επίσης χαιρόμαστε που στον πρώτο πυλώνα συμπεριλήφθηκε το πρασίνισμα και υπάρχει και η κατανομή η ισότιμη και ισόρροπη των άμεσων ενισχύσεων για τις 27 χώρες. Πρώτη φορά έχουμε ένα φθήνον σύστημα ε, ενισχύσεων βάσει κριτηρίων που έχουν να κάνουν με την απασχόληση και με το περιβάλλον. Πρέπει να θαρρύνουμε τους νέους αγρότες που αναλαμβάνουν ε, νέα καθήκοντα κοντά στη γη, στην Ήπεθρο και να φροντίσουμε επίσης να προστατεύσουμε περισσότερο το περιβάλλον το οποίο τόσο πολύ χρειαζόμαστε. Κυρία Σάρμπου, τώρα για ένα λεπτό. Κύριε Επίτροπε, χρειαζόμαστε μία γεωργία που να διασφαλίζεται από μία ΚΑΠ με κατάλληλο προϋπολογισμό. Έτσι θα προστατεύσουμε και ε, τα τρόφιμα από οποιαδήποτε κρίση. Και θα δώσουμε και τα κατάλληλα εισοδήματα στους αγρότες για να ζουν αξιοπρεπώς. Αυτή πρέπει να είναι και η βάση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Είναι λάθος να μιλάμε για περισσότερη συνέχεια στις άμεσες πληρωμές μεταξύ των γεωργών και των χωρών. Αν υπάρχουν διαφορές, αδικαιολόγητες πρέπει να καταργηθούν. Σημειώνω και την πρόταση της Επιτροπής για απλοποιημένο πρόγραμμα όσον αφορά τις μικρές εκμεταλλεύσεις. Τα προγράμματα για τους νέους γεωργούς είναι επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει να υποστηρίξουμε για να συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη της υπαίθρου και να διασφαλίσουμε ότι οι νέες γενιές θα συνεχίσουν να απασχολούνται στη Γεωργία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σάρμπου. Εδώ τελείωσαν οι παρεμβάσει των βουλευτών, εγγεγραμμένων βουλευτών και ερχόμαστε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye. Ενδιαφέρον θέμα, έχουν ζητήσει το λόγο πολλοί συνάδελφοι. Δεν θα τον πάρουν όλοι. Ε, θα κρατήσω τη σειρά που τον ζήτησαν. Ε, θα δώσω το λόγο καταρχάς στην κυρία Αντωνέσκου. Ένα λεπτό παρακαλώ, μην το ξεπεράσετε για να μπορέσουν να πάρουν το λόγο στον το περισσότεροι. Η κυρία Αντωνέσκου για ένα λεπτό. Λοιπόν, η κυρία Αντωνέσκου δεν, μπόρεσε να περιμένει μέχρι το τέλος. Ο κύριος Καλίνοφσκι για ένα λεπτό παρακαλώ. Dziękuję bardzo, Πρόεδρε, κύριε πίτροπε, κατά τη γνώμη μου, η έκθεση DES έχει ένα μεγάλο ελάττωμα, ελάττωμα στο σημείο 16. Αυτό έρχεται σε αντίθεση, αυτό σημείο, με την βασική αρχή του, της αρχής του ανταγωνισμού στην κοινή αγορά. Ε, δίκαιος ανταγωνισμός στην κοινή αγορά. Υπάρχουν ε, διαφορές στις άμεσες πληρωμές για τους γεωργούς στα διάφορα κράτη-μέλη. Κάποιοι θα παίρνουν 200-250 ε, ευρώ ανεκτάριο, άλλοι 350-400 ε, ευρώ. Αυτό δεν εξασφαλίζει την ισότητα μεταξύ των μικρών και των μεγάλων κρατών μελών, των παλιών και των νέων κρατών μελών. θα πρέπει να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για τον ανταγωνισμό στη γεωργία. Φυσικά υπάρχουν διαφορές, αλλά θα πρέπει να απορρέουν μόνο από αντικειμενικά κριτήρια. τώρα θα πάρει το λόγο ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η σημασία της ε, ΚΑΠ και του ρόλου που παίζει για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την ε, διατροφική ασφάλεια είναι γνωστή σε όλους. Οι περιβαλλοντικές ε, προκλήσεις, ε, η καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής καθιστούν την ΚΑΠ μετά το 2013 ακόμα πιο σημαντική. Θα πρέπει να είναι πιο ισχυρή, πιο βιώσιμη και θα πρέπει να έχει μια πρικοδότηση από τον προϋπολογισμό ικανοποιητική για να μπορέσει να υλοποιήσει τους ε, στόχους που έχουμε θέσει με μια ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη προϊόντων ε, διατροφικών ποιοτικών και να εξασφαλίσει τις ανάγκες των μικρών γεωργών η κερδοφορία, κερδοσκοπία στις πρώτες ύλε και η φοβερή ε, αστάθεια των τιμών ε, διακυβεύουν την διατροφική ασφάλεια και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε ε, ευέλικτα μέσα. Μπορεί, θα πρέπει να έχουμε αντικυκλικά μέτρα για να αντιμετωπίσουμε τις αλλαγές στην αγορά. όλα αυτά στον πρώτο πυλώνα για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε έγκαιρα και αυτόματα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή δεν δίνει απαντήσεις στις προκλήσεις, τις μελλοντικέ που έχουμε και που προβλέπονται και από τον τίτλο στο κάτω-κάτω. Δεν καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε ούτε τα σημερινά προβλήματα. Γι' αυτό και εμείς υποβάλλουμε τροπολογίες που πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίες προκειμένου να τροποποιηθεί σε βάθος η σημερινή ΚΑΠ. Θέλω να υπογραμμίσω εδώ τα δύο μέσα ρύθμισης των αγορών και τους μηχανισμούς παρέμβασης που πρέπει να διασφαλίσουν καλές τιμές για τους αγρότες και έτσι να μπορούν όλες οι χώρες να έχουν το δικαίωμα να παράγουν. Το ίδιο σκύει και για τις ποσοστώσεις γαλακτοκομικών προϊόντων προκειμένου να στηρίξουμε τους παραγωγούς των πιο ευάλωτων χωρών. Θέλουμε επίσης να διατηρηθούν και οι ενισχύσεις για να αντιμετωπίζονται οι κρίσεις που προκύπτουν. Επίσης να προβλέπονται και κάποιες ενισχύσεις σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Θέλουμε μια γεωργία που να προστατεύει το περιβάλλον. Μερικές φορές όμως αυτό δεν γίνεται με τη σημερινή αγορά όπως έχει. Κύριε συνάδελφοι, στερείτε το λόγο από άλλους συναδέλφους. Ο κύριος Ρώση. δεν είναι εδώ. Ε, το λόγο τώρα θα πάρει η κυρία... Θα πάρει ο κύριος Μπρόνς. Συγγνώμη, ο κύριος Μπρόνς. Uh, Εμείς θέλουμε να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και επομένω δεν θέλουμε και την ΚΑΠ. Ε, όμως αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να τη μετωπίσουμε. Ε, τι, άποψη έχουμε για την έκθεση ΔΕΣ. κάποια τμήματα είναι καλά. Το να δώσουμε άμεσες πληρωμές και αυτό να εξαρτάται από τη διασταυρούμενη συμμόρφωση για θέματα περιβάλλοντος και την διαφύλαξη της υπαίθρου, ίσως αυτό είναι ευεργετικό ενδυνάμει ευεργετικών, μόνο εφόσον δεν συνδέεται από κάποιες, έτσι, από αυτά τα θέσφατα που έχουμε θέσει για την κλιματική αλλαγή κτλ. Η έκθεση αναγνωρίζει ότι ο γεωργικό τομέα θα πρέπει να εξακολουθήσει να υποστηρίζεται από κυβερνητικέ επιδοτήσει. Γιατί ούτω ή άλλω δεν μπορούμε να προβλέψουμε ακριβώ ε, τι καλλιέργειε και η δεν μπορούμε να ξέρουμε τη ζήτηση που θα έχουν τα γεωργικά προϊόντα. Αυτό είναι σημαντικό. Επίσης είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ε, την διατροφική ασφάλεια και να αποφύγουμε την αστάθεια των τιμών. Το πιο σημαντικό, κάτι, την άποψή μου, είναι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να σταματήσει να είναι ε, σημαντικός ε, πληρω, πληρωτής της ΚΑΠ. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η δουλειά αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική που έγινε από τον εισηγητή. Έχουμε καταλήξει σε ένα έγγραφο ισορροπημένο για την ΚΑΠ. Είναι ένας καλός προσανατολισμός για τις νομοθετικές προτάσεις που θα ακολουθήσουν. Γι' αυτό και συγχαρητήρια στον εισηγητή. Έχω όμως κάποιες, μάλλον, κάποιες από τις προτάσεις που περιλαμβάνονται εδώ με ανησυχούν κάπως και θα παρακολουθήσω τι θα γίνει στη συνέχεια. Για παράδειγμα, η κατανομή ενισχύσεων του πρώτου πυλώνα. Πρέπει να βασιζόμαστε σε αντικειμενικά κριτήρια. Το κριτήριο της κατανομής δηλαδή να μην αλλάζει και γίνεται συνοχής όπως είναι σήμερα. Χρειαζόμαστε μια πιο δίκαια ΚΑΠ με έναν κατάλληλο προϋπολογισμό. Πρέπει επίσης να επιβεβαιώσουμε την ανάγκη ότι ο αλλακτοκομικός τομέας θα συμπεριληφθεί στην ατζέντα με την έγκριση των τροπολογιών 16, 12 και 5. Όλοι ναι, τσακ έχει το λόγο. Ένα λεπτό παρακαλώ. Celem wspólnej polityki rolnej jest zagwarantowanie ciągłości w dostarczaniu żywności dla mieszkańców Europy. I ΚΑΠ στόχο έχει να δώσει τρόφιμα στις ευρωπαϊκές αγορές. Θα πρέπει να δώσουμε τρόφιμα α, υψηλής σε προσιτές τιμές. Αυτό περιμένουν οι καταναλωτές. Ε, με την παραγωγή και την ε, μεταποίηση θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και την προστασία του περιβάλλοντος. Είμαστε υπέρ της ΚΑΠ, αλλά δεν θέλουμε να επανεθνικοποιηθεί η γεωργία. Θέλουμε μεγάλο προπολογισμό, δεν θέλουμε περικοπές. Οι άμεσες πληρωμές θα πρέπει να δοθούν με απλό τρόπο ισότιμα σε όλους τους γεωργούς, σε όλες τις χώρες. Ε, θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι άμεσες πληρωμές είναι μόνο τμήμα του εισοδήματο των αγροτών. Επομένως, θα πρέπει να υπάρχει ρύθμιση της αγοράς, κατάλληλες τιμές και σταθερότητα στην αγορά. Όλα αυτά εξασφαλίζουν το δίκαιο εισόδημα των ε, γεωργών. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε στους κατοίκους της ε, υπαίθρου ότι έχουν πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, ε, μεταφορές, υγεία, εκπαίδευση, αθλητισμός και πολιτισμός. Αυτό θα πρέπει να υπάρχει στο δεύτερο πυλώνα και στην πολιτική συνοχής. Ε, Κομισιόν. Αφήστε μας να διατηρήσουμε ε, το πρόγραμμα που βάζει επίσης ε, φαγητό στο πιάτο των, φτωχών. Una Σχετικά με τη διατροφική ασφάλεια, η ΚΑΠ πρέπει να απαντήσει σε αυτή την πρόκληση και η νέα πολιτική θα πρέπει να συνεχίσει τα θετικά στοιχεία της παρούσης και να διορθώσει τα λάθη. Μας προτείνουν ε, δύο πυλώνες, τις άμεσες πληρωμές και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Πρέπει όμως να υπάρξουν ε, αντικειμενικά κριτήρια. Δεν είναι είναι ίσες οι άμεσες πληρωμές για όλα τα κράτη-μέλη αλλά πρέπει να είναι λογικές οι διαφορές λαμβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές και κοινωνικές διαφορές με ένα κατώτατο και ανώτατο ε, πλαφόν ε, για τον μέσο όρο της Ευρώπης για να μπορέσει να προωθηθεί και οικολογικά ένας προπολογισμό της Ευρώπης ίσως με αυτόν τον ο οποίος θα ισχύσει το 2013. Αυτό που μας χαροποιεί είναι ότι η πρώτη έκθεση του Κοινοβουλίου έχει πολλά κοινά. Ο Ευχαριστώ. Το πιο σημαντικό μήνυμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα είναι ότι θέλει μια δίκαια ΚΑΠ. Δηλαδή μια ΚΑΠ η οποία να διασφαλίζει επαρκή έσοδα για όλους τους παραγωγούς. Όπου και αν ε, ζουν, όπου και αν ε, δουλεύουν, ό,τι και αν παράγουν. Άρα λοιπόν οι άμεσες ενισχύσεις έχουν πολύ μεγάλη σημασία γιατί στηρίζουν και την ανάπτυξη τη υπαίθρου και φροντίζουν να ανταποκριθεί η ΚΑΠ στη στρατηγική του 2020. Πρέπει όμως να σέβεται τους περιβαλλοντικούς και άλλους στόχους που έχουμε θέσει. Χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτό που είπε ο Επίτροπος, ότι δηλαδή στον πρώτο πυλώνα θα δει και όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν για την εγκατάσταση νέων στις αγροτικέ δραστηριότητες. Είναι πολύ σημαντικό να βρούνε καλές συνθήκες στην ε, διαβούλευση πρέπει να φροντίσουμε να τους ακούσουμε για να μπορέσουν να βρεθούν περισσότεροι αγρότες στην Ήπεθρο. Υπάρχουν χώρες οι οποίες στηρίζουν τους νέους αγρότες. Αυτούς ε, που δεν κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν τις δραστηριότητε τους, αλλού όμως όχι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντως πρέπει να φροντίσει να ενισχύσει αυτούς και να μην βασίζονται μόνο στην εθνική πολιτική. Thank you Ευχαριστώ. Président. Κύριε Ταταρέλα, δεν είμαι ο κύριος Ταταρέλα, είμαι ο κύριο Ταραμπέλα, αλλά δεν με προσβάλετε. Ε, διαδικαστικό, θέλω να σας πω. Σκανδαλώδης στάση της ε, Ουγγρικής ε, Προεδρίας, που είναι μία από τις χειρότερες που έχουμε δει ποτέ ε, η οποία παρέστη στην πρώτη συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, βγήκε τώρα για τα γεωργικά και τώρα ξαναμπαίνει για την οικονομική διακυβέρνηση. Βλέπετε τι σημασία δίνει στην Ευρωπαϊκή Γεωργία και στους γεωργούς της Ευρώπης. Είναι το 40% του, του προπολογισμού. Καλό θα ήταν η Ουγγρική Προεδρία να είχε κάτσει να ακούσει τη συζήτηση. Αυτό ήθελα να πω, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Elnézést kérek, hogy a de most Ευχαριστώ. Μόλις έφτασα, δεν ξέρω τι έχει διαμειφθεί μέχρι στιγμής, αλλά τώρα ο κύριος Ντερόση έχει τον λόγο, δεν είναι όμως εδώ. Ευχαριστώ. Είμαστε υπέρ αυτή τη έκθεση πρωτοβουλία. Γιατί η ΚΑΠ είναι το βασικό εργαλείο για την Ευρωπαϊκή Γεωργία και για την προστασία των παραγωγών των προϊόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στα ξένα προϊόντα. Τα βασικά στοιχεία τη έκθεση είναι η διατήρηση των δημοσιονομικών στοιχείων, νέα κριτήρια κατανομής, ε, πώς μπορούμε να τα δεχτούμε. Εγκαταλείπεται το κριτήριο, το ιστορικό όμως, ως παράμετρος για τη διανομή των άμεσων πληρωμών προβλέπονται ε, πρημοδοτήσει τη ε, εκμεταλλεύση. Λαμβάνεται υπόψη ε, η εργασία και το κόστο τη παραγωγή. Απλουστεύεται ο τρόπο πληρωμή. Ζητάμε οι άμεσε πληρωμέ να δίδονται μόνο στου ενεργού γεωργού και να υπάρχουν και ανώτατα όρια. Ούτω ώστε οι αποδέκτε να είναι αυτοί που πραγματικά καλλιεργούν τη γη και όχι οι κερδοσκόποι. Άλλο σημαντικό σημείο, κατά την άποψή μα, είναι η ανάπτυξη υπαίθρου η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που έχουμε ε, στο έδαφος και στους ανθρώπινου πόρου, προστασία των ε, ορεινών περιοχών. Η νέα ΚΑΠ θα πρέπει μεταξύ των στόχων τη να έχει ε, την ένταξη των νέων διοργών, κυρίως των νέων, με συγκεκριμένα συγκεκριμένε πιστώσει χρηματοδότηση, να μειωθεί επίση και το κόστο και η γραφειοκρατία για αυτού. Με συγχωρείτε, διότι Υπάρχουν 20 άτομα στη διαδικασία Catch the Eye, αλλά θα δώσω το λόγο μόνο σε 10. Ο κύριος Ντόρφμαν έχει τώρα το λόγο για ένα λεπτό και θα είναι ο τελευταίος ομιλητής. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, με την έκθεση DES ε, προβαίνουμε σε ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για την γεωργική πολιτική και είναι βασικό να υπάρξει μία σωστή αιτιολόγηση για την κατανομή των ε, χρηματοδοτήσεων. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει η κατανομή πόρων στον πρώτο πυλώνα να είναι πιο δίκαια και θα πρέπει να ανατρέξουμε και στις ιστορικές πολλές Υπάρχουν πολλοί τρόποι κατανομής μεταξύ κρατών μελών αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε και για την κατανομή εντός των κρατών μελών που υπάρχουν μεγάλες ανισότητες όπου αλλού πρέπει να εξετάσουμε περισσότερο και να βοηθήσουμε τις μικρότερες επιχειρήσεις. Επίσης έγινε μία έκθεση για μία νέα οριοθέτηση. Δεν ακούσαμε τίποτα περαιτέρω θα ήθελα να ξέρω τι σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του θέματος αυτού. Ευχαριστώ. Κύριος Τσιόλος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είχαμε μια συζήτηση μια ώρας για την έκθεση DES και είμαι πολύ αισιόδοξο. όχι μόνο για την ψηφοφορία που θα λάβει χώρα αύριο και για το αποτέλεσμα της έκθεσης που όπως είπα και στην αρχή μοιάζει πολύ με αυτά που πρότεινε η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς, αλλά είμαι πολύ αισιόδοξο και για το μέλλον της κοινή μας γεωργικής πολιτικής επαναλαμβάνω, όπως είπα και στην αρχή, το ότι είμαι πιστός στην αρχή μου ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία και συμπληρωματικότητα ανάμεσα στους δύο πυλώνες της κοινή γεωργικής πολιτικής. Και η μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική πρέπει να συνεχίσει να έχει ένα δεύτερο πυλώνα ισχυρό, γιατί έχουμε πολλές φιλοδοξίες για το δεύτερο αυτό πυλώνα, για την ισορροπία δηλαδή μέσα στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια για τη στήριξη της μικρής γεωργίας των νέων γεωργών και την ανάπτυξη της υπαίθρου μας. Σας διαβεβαιώνω λοιπόν και εγώ και ο πρόεδρος Μπαρόσο και ολόκληρη η Επιτροπή δίνει μεγάλη σημασία στο δεύτερο πυλόν, ο οποίος δεν πρόκειται να πληρώσει το τίμημα ε, τη συζήτηση για τον καινούριο κοινοτικό προπολογισμό. Σα το λέω και σα το λέω και εκ μέρου του Πρόεδρου Μπαρόσο. Στη συνέχεια, δεν θα ήθελα και εξάλλου η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της δεν βάζει σε αντίφαση το θέμα της παραγωγής τροφίμων με ε, το θέμα του περιβάλλοντος. Αυτό το οποίο προτείνουμε είναι ισορροπία ώστε από τη μια μεριά η οικονομική ανταγωνιστικότητα και από την άλλη μεριά η προστασία των φυσικών μας πόρων να προχωρήσει. Γιατί δεν γίνεται αλλιώ. Χρειάζεται ισορροπία μεταξύ των δύο. Πρέπει να προσέξουμε και τους φυσικούς πόρους. Δεν πρέπει άρα να βάλουμε σε αντίθεση το θέμα της παραγωγής τροφίμων με το θέμα του περιβάλλοντος στη μελλοντική ΚΑΠ. Έπειτα, να στοχεύσουμε καλύτερα τα θέματα μας. Ο κύριος Άσφουλτ το έθεσε, αλλά δεν βλέπω να είναι εδώ πια. Σε αυτά που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στοχεύουμε πολύ καλύτερα το θέμα των άμεσων πληρωμών. Και αυτό είναι που προτείνει και ο κύριος ε, Ντες στο κάτω-κάτω. Ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τις προτάσεις που θα κάνει τις νομοθετικές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έρχομαι τώρα στην κρίση. Θα υπάρξουν μέτρα ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και στο μέλλον κρίσεις που έχουν να κάνουν με την κατάσταση στην αγορά, που είναι ε, θέματα υγιεινής ή οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο για την στήριξή του προκειμένου οι ακρότες μας να μπορέσουν να είναι ήσυχοι όσον αφορά το μέλλον. Θα ολοκληρώσω εκφράζοντας για άλλη μια φορά την αισιοδοξία μου όσον αφορά την αυριανή ψηφοφορία και όσον αφορά την έκθεση ΔΕΣ. Σας ε, διαβεβαιώνω τον Οκτώβριο στο πακέτο νομοθετικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα βρείτε όλα τα βασικά στοιχεία που περιλαμβάνει η έκθεσή σας. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ πολύ για την δουλειά σας που αποτελεί μια πρόσθετη αξία στο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Και τώρα Κλείνοντας αυτή τη συζήτηση, δίνουμε το λόγο στον εισηγητή, στον Άλμπερτ Ντέσσα. Κύριε Πρόεδρε, <clears throat> κύριε Επίτροπε, αγαπητές κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για το πνεύμα της συζήτησης και για την στήριξη που μας δόθηκε. Κύριε ε, Επίτροπε, προσβλέπουμε όλοι στην ανακοίνωσή σας τον Οκτώβριο και στη συνεργασία, διότι η Γεωργία τρέφει πάνω από 550 εκατομμύρια άτομα τεράστια τις εκτάσεις ε, σε απόμακρες περιοχές ε, και είναι βασικός χώρος της υπαίθρου και έχουμε μία βιώσιμη γεωργία. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί ο πρόεδρος Μπαρόζο μίλησε για σημαντικές περικοπές στον δεύτερο πυλώνα διότι έτσι θέτει σε κίνδυνο και τους στόχους του 2020, τους δικούς του ε, ε, τους δικούς τους στόχους. αν ε, 15 εκατομμύρια γεωργοί τρέφουν 50 εκατομμύρια άτομα τότε θα πρέπει να αναφέρουμε 500 εκατομμύρια άτομα πρέπει να πούμε ότι εγώ είμαι μεν πολύ καιρό πολιτικός και ξέρω γιατί διατύπωσα έτσι την έκθεσή μου. Εάν είχε σήμερα ε, αν είχε η έκθεσή μου αρχικά την εικόνα που έχει τώρα τότε δεν θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε συμβασμούς και να έχουμε μία αίσια έκβαση σαν αυτή που επιτύχαμε. Θέλω λοιπόν να επιτύχω να δώσουμε ένα σήμα σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι εξετάζουμε τα πιο βασικά θέματα που είναι βασικά τα οποία εξασφαλίζουν ένα καλό μέλλον για τους γεωργούς και τις οικογένειές τους και θα πρέπει όλοι να συνεργαστούμε κύριε Επίτροπε για να επιτύχουμε το στέχο αυτό και θέλω να σας πω ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχετε περισσότερο περισσότερη στήριξη από ότι άλλοι επίτροποι και αυτό μπορούμε να σας το εξασφαλίσουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Ντές. Ε, με αυτό κλείνει το σημείο στη συζήτηση.